possiamo iniziare i lavori Ξεκινάμε εκ νέου λοιπόν τις εργασίες της Επιτροπής μας. Ελπίζω να πάμε νωρίς στην αρχή. Να πάμε γρήγορα, συγγνώμη, στην αρχή. Έχετε νομίζω όλοι το σχέδιο ημερησίας διάταξης. Έχετε παρατηρήσεις, όχι. Θεωρείται δεκτό λοιπόν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Το δεύτερο σημείο αφορά την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας την 1η και τη η Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ε, των συντονιστών υπήρξε μια παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα και η κυρία Γκρινή θα σας παρουσιάσει την αίτηση τροποποίηση των πρακτικών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι στα πρακτικά λέγεται ότι θα υπάρξει μια επίσκεψη στη Μαδρίτη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της τελευταίας δεν μιλήσαμε εμείς για Μαδρίτη. Εμείς μιλήσαμε μόνο για επισκέψεις στην Αυστρία και στην πόλη Χουέλβα της Ισπανίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διορθωθούν παρακαλώ τα πρακτικά. Καλώς δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν θα γίνει αυτή η διόρθωση στα πρακτικά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. με τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η κυρία Παλιαδέλη Σιγήτρια Και επόμενο θέμα, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την δραστηριότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με γνωμοδότρια την κυρία Άουκεν. Η κυρία Άουκεν δεν είναι παρούσα για προσωπικούς λόγους και δεν θα μπορέσει φυσικά να πάρει το λόγο αλλά νομίζω ότι μιας και δεν έχουν υπάρξει τροπολογίες και γι' αυτό νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη εκτός αν κάποιος από εσά έχει διαφορετική άποψη. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Παλιαδέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Ομολογώ ότι όταν μου ανατέθηκε αυτή η ευθύνη για να κάνω την πρώτη μου εισήγηση εδώ στην ε, Επιτροπή Αναφορών ε, για έναν τόσο σημαντικό θεσμό όπως είναι ο θεσμός του Ευρωπαίου Μεσολαβητή ένιωσα λίγο περίεργα αν θα τα καταφέρω. Διαπίστωσα όμως τις εξαιρετικές ικανότητες ε, ολόκληρης της γραμματείας του κυρίου David Λόου και βεβαίως της κυρίας Κάριν Χιώτη στους οποίους πολλό, ε, ομολογώ ότι πρέπει να ζητήσω να δώσω μεγάλη, πολλά ευχαριστώ για την βοήθεια και για τις παρατηρήσεις τους ο άλλος λόγος για τον οποίο θα ένιωσα ε, περίεργα όταν ανέλαβα αυτή την αναφορά ήταν ε, η σπουδαιότητα του θεσμού αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο, ο, ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής, ο κύριος Διαμαντούρος. Και αυτό γίνεται φανερό όχι μόνο από ε, τη μορφή των εντύπων τα οποία είχατε στη διάθεσή σας όχι μόνο την αναλυτική έκθεση αλλά και την σύντομη επισκόπηση αυτής της έκθεσης από την οποία προκύπτουν, προκύπτει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο Ευρωπαίος ε, διαμεσολαβητής το καθήκον του, ε, τις, ευθύνες του με επίκεντρο τον Ευρωπαίο πολίτη. Και από την άποψη αυτή νομίζω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα ότι υπάγομαι σε μια επιτροπή που και αυτή έχει μια άμεση σχέση με τον Ευρωπαίο πολίτη. Διαβάσατε φαντάζομαι την έκθεση, διαβάσατε επίσης και την αιτιολογική έκθεση. Θα ήθελα να πάρω πολύ σύντομα λίγο από τον χρόνο σας. Ε, μιλώντας για αυτήν, θεωρώ ότι πολύ σημαντικός και πολύ φιλικός προς, το, προς τον αναγνώστη και τον χρήστη είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή τα στατιστικά δεδομένα, ε, οι αριθμοί δηλαδή με τους οποίους βρέθηκε αντιμέτωπο στη διάρκεια ενός χρόνου ο διαμεσολαβητής και το γραφείο του. 3.406 ε, καταγγελίες στη διάρκεια του χρόνου που μας πέρασε, ε, από τις οποίες 802 ήταν εντός των πλαισίων των ε, ε, δικαιοδοσιών και των υποχρεώσεων του διαμεσολαβητή. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένα μεγάλο ποσοστό, το 36% των περιπτώσεων, αναφέρεται σε ε, κακοδιαχείριση που σχετίζεται με την έλλειψη της διαφάνειας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαπίστωση ε, για όλους μας. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ο τρόπος με τον οποίο, οι τρόποι μάλλον με τους οποίους ο ε, διαμεσολαβητής και το γραφείο του διεκπαιρέωσαν ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές. Μια προσπάθεια για έναν φιλικό διακανονισμό θα λέγαμε ανάμεσα στον ε, καταγγέλλοντα και στον φορέα ή τον θεσμό με προς τον οποίο αναπευθυνόταν η καταγγελία. Πέρα από αυτή την πρόταση, από αυτή την μέθοδο, ε, ο διαμεσολαβητής έδειξε και την ε, ισχύ με την, τη διάθεση να λύσει τα ζητήματα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπος με τις επικριτικές του παρατηρήσεις. Ε, μιας, ε, μια, μια μέθοδο η οποία οδήγησε τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν διορθωτικές επεμβάσεις στις υποθέσεις για τους οποίους είχαν καταγγελίες. Είναι ενδιαφέρον ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής συμβουλεύτηκε τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή άλλους φορείς που σημαίνει μια διάθεση από τη μεριά του για συνεργασία ε, προκειμένου να απαντηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η καταγγελία. Πέρα από αυτό θα ήθελα να τονίσω τις δύο μελέτες που δημοσιεύτηκαν στη διάρκεια του 2008 και αφορούσαν γενικότερα ζητήματα που σχετίζονται με επικριτικές παρατηρήσεις του 2006 και του 2007. Εντός του 2008 ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής υπέβαλε και 8 σχέδια συστάσεων προς, προς τους ε, θεσμούς ή τους φορείς με τους οποίους υπήρχε το πρόβλημα, ενώ ε, το 2008 ο ίδιος κατέθεσε ειδική έκθεση επικρίνοντας την Επιτροπή ότι δεν αξιολογεί, δεν αιτιολογεί επαρκώς τη συμπεριφορά ε, σε ορισμένους τομείς όπως είναι η επικουρική διερμηνής. Ε, ένα άλλο ζήτημα με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπος και το οποίο θεωρώ εξαιρετικής ευαισθησίας είναι η αυτεπάγγελτη έρευνα που αφορά στις καθυστερημένες πληρωμές ε, ορισμένων προμηθευτών της Επιτροπής. Ζήτησε από την Επιτροπή να υπάρξουν βελτιώσεις περισσότερες από αυτές που αρχικά ε, προτάθηκαν και βεβαίως ε, έλαβε την υπόσχεση ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί εντός του 2009. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο διαμεσολαβητής ανακοίνωσε πως σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο θα ξεκινήσει νέα έρευνα. Ε, θα, έκλει, θα κλείσω αυτή την σύντομη παρουσίαση σε, ε, με τις προτεραιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που στην ουσία ταυτίζονται απόλυτα με τις προτεραιότητες όλων μας σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τους Ευρωπαίους πολίτες, το σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών σε κάθε επίπεδο, τη βελτίωση της ποιότητας της ενημέρωσης, κάτι που ήδη έχει γίνει με αυτά τα κομψά κείμενα και με την ιστοσελίδα, και βεβαίως την ε, έκκληση προς τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής, Έρευνας, ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν μια τακτική που θα λύνει τα προβλήματα ή που θα αντιμετωπίσει τον πολίτη με το δέοντα σεβασμό και θα ενθαρρύνει τη βέλτιστη πρακτική. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα κατά συνέπεια ότι για τους παραπάνω λόγους ε, θεωρώ ότι η έκθεση αυτή όπως κατατέθηκε γραπτά και όπως υλοποιείται ε, μορφικά με τη σύντομη επισκόπηση και με την ετήσια μορφή της εγκρίνεται θα λέγαμε ότι γίνεται αποδεκτή από τον εισηγητή γιατί καλύπτει απολύτως βασικές αρχές της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιώντα μια πρόθεση να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, ένα βασικό αιτούμενο, να περιφρουρήσει τη διαφάνεια και να προωθήσει ένα πνεύμα εξυπηρέτηση των πολιτών που θα ενθαρρύνει την ε, τάση τους να λύνουν ζητήματα που τους αφορούν μέσω του Ευρωπαίου Μεσολαβητή. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι ότι έπεσα την ώρα που προσφέρετε καφές, αλλά ελπίζω ότι ακούσατε όλα αυτά που είχα να σας πω. Αν δεν θέλει κανείς ε, το λόγο, έχουμε τροπολογίες για την έκθεση, θα τις ψηφίσουμε, αλλά το λόγο ζήτησε η κυρία Γκρουνή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Παλιαδέλη ε, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζουμε πλήρως την πρόταση της ε, κυρίας Παλιαδέλη, την οποία και συγχαίρουμε. Εν μέρη υποστηρίζουμε τις τροπολογίες ε, της κυρίας Κοχμέριν, όχι όλες. Λίγες τροπολογίες έχουμε, κυρίως συντακτική φύσεως, οπότε δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Απλώς απορρίπτουμε την πρώτη προφορική τροπολογία των πρασίνων και για τη διαδικασία λίγο να θυμίσουμε ε, τις προθεσμίες για τις μεταφράσεις των εκθέσεων στις γλώσσες μας γιατί είναι δύσκολο για τις τροπολογίες να δράσουμε χωρίς να τις έχουμε μεταφρασμένες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, την κυρία Γκρινή, πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα και όσο πληθαίνουν οι γλώσσες τόσο θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Ε, αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε χρόνο ομολογουμένως ούτε για περισσότερες τροπολογίες και αυτό πρέπει να το πούμε γιατί κατατέθηκε στις 21 Απριλίου και έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει η διαδικασία. Ελπίζουμε ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά οι τροπολογίες ήταν ε, λίγες σχετικά και ευχαριστώ τους συναδέλφους. Είναι συνολικά 17 τροπολογίες και δύο προφορικές τροπολογίες. Ε, ήδη έχουμε την άποψη της, ε, του ΕΠΠ. Δεν ξέρω αν έχουμε και ε, Ευχαριστώ κυρία Παλιαδέλη. Άλλε πολιτικέ ομάδε θέλουν το λόγο. Οπότε α περάσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτη τροπολογία τη κυρία Παλιαδέλη στην παράγραφο 3. Στην αιτιολογική αναφορά μάλλον 3. Σιτασιόν 3. Αιτιολογική αναφορά. Favorevoli υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 της κυρίας Παλιαδέλης, το G, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία. Παράγραφος πρώτη. της κυρίας Κοχμερίν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 2. Πάλι Κοχμερίν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Παράγραφος 5. Πάλι Κοχμερίν. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει καταδιέρεση ψηφοφορίας. Θέτω σε ψηφοφορία το πρώτο τμήμα. Μέχρι εκεί που λέει και με διαφάνεια. Βέβαια στις διάφορες γλώσσες είναι γραμμένο με διαφορετικό τρόπο. και είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή η τροπολογία. Το δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Στην παράγραφο 5 τελευταία φράση η τροπολογία της κυρίας Παλιαδέλη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στην παράγραφο 6. Προφορική τροπολογία της κυρίας Άουκεν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία Κοχμερίν. Και εδώ θα γίνει κατά διέρεση ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Θέτω σε ψηφοφορία λοιπόν το πρώτο τμήμα της νέας διατύπωσης. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Θεωρεί όμως και μετά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Η τροπολογία της κυρίας Παλιαδέλη και της κυρίας Ράπτη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 9. Τροπολογία της κυρίας Κοχμερίν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 10. Τροπολογία της κυρίας Παλιαδέλη. Είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 10 πάντα. Τροπολογία της κυρίας Κοχμερίν. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαναλαμβάνουμε ποιοι είναι υπέρ. Κατά. δεκτή, δεκτό το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα τώρα δεν θα ψηφιστεί εφόσον έχει γίνει δεκτό το πρώτο. Στην παράγραφο 11, τροπολογία της κυρίας Παλιαδέλη, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στην παράγραφο 16, προφορική τροπολογία Άουκεν. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές δεκτή. Στην παράγραφο 20 τροπολογία Κοχμερίν είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στην παράγραφο 20 της κυρίας Παλιαδέλη είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στην παράγραφο 22 πάντα της κυρίας Παλιαδέλη ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Στην παράγραφο 23 της κυρίας Παλιαδέλη υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Στην παράγραφο 23 της κυρίας Κοχ σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα έχει καταπέσει πλέον. Τελική ψήφος για το σύνολο της εκθέσεως, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, η έκθεση γίνεται δεκτή. Βλέπω ότι ήρθε η κυρία Άουκεν. Οπότε μπορούμε να πάμε στο σημείο 8. για την ψηφοφορία. για το θέμα στο οποίο είναι η συγγήτρια η κυρία Ούκεν. Δεν υπάρχουν τροπολογίες όπως σας είχα πει και στην αρχή, οπότε περνάμε απευθεία στις ψηφοφορίες. Άρχεται η ψηφοφορία, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά τις ψηφοφορίες θα περάσουμε τώρα στην εξέταση ορισμένων αναφορών πλέον σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τους φυσικούς οικοτόπους. Πριν από την εξέταση αυτής, ε, αυτών των αναφορών θα ακούσουμε έναν από τους ε, συγκαταθέτες αυτών των αναφορών. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα ίσως Ένας από αυτούς λοιπόν που έχουν συγγράψει την έκθεση που έχουμε στην ημέρηση αδιάταξη. το είχαμε πει και στην τελευταία συνεδρίασή μας υπάρχουν αρκετές αναφορές οι οποίες είναι γύρω από το ίδιο θέμα και θα μας απασχολήσουν σήμερα το πρωί. Για τις αναφορές αυτές σήμερα το πρωί έχουμε παρόντες αυτούς που έχουν καταθέσει την οδηγία 12 ο κύριος Ζαμαρή Σαλωμό 13 ο κύριος Νταβίτ Κολόν και ο Ζαν Πολ Ντεκλέρκ. Σχετικά στην αναφορά 15 ο Μάρκ Βεσάουερ δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα, αλλά θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον σχετικά με την αναφορά 15. Ελπίζω να λύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα. Allora, mentre risolvono i problemi Πόσο λύνονται τα τεχνικά θέματα θα σας δώσω κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Ξέρετε ότι στα τελευταία πρακτικά είναι οι αναφορές οι οποίες γίνονται αποδεκτές, είχαν γίνει αποδεκτές μάλλον. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο ή αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Αν δεν κάνετε παρατηρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης θεωρείτε δεκτό. την προηγούμενη εβδομάδα μοιράστηκε σε κάποιους από εσά, σε όλους σας μάλλον, ο κατάλογος των αναφορών που θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση για τον κατάλογο αυτό, θα πρέπει να θεωρηθεί δεκτός. αν και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τη 0704 του 2008, εδώ θα ήθελα να ζητήσω περισσότερο χρόνο, θα πρέπει να επανέλθουμε. Σχετικά με το δεύτερο τμήμα του εγγράφου, όπως γνωρίζετε ήδη, και εφόσον δεν υπάρχουν σχόλια και αντιρρήσεις, το δεύτερο αυτό τμήμα σαν πρόταση θεωρείται δεκτό. Θέλει κάποιος να κάνει σχόλια για το δεύτερο τμήμα. Όχι. Οπότε εγώ πάλι θα πάρω το λόγο και θα ζητήσω να σταματήσει η αξιολόγηση του 53, 52 και 56 προσωρινά. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για το σημείο 82. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Θεωρείται δεκτή η πρόταση. Καλώς. Κλείνουμε λοιπόν και η τελευταία ανακοίνωση αφορά τη σημερινή συνεδρίαση των συντονιστών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών διακόπτη πρόεδρος. Στα πλαίσια λοιπόν της συνεδρίασης των συντονιστών θα σας ενημερώσω ότι συμφωνήθηκε να ξεκινήσουμε την εξέταση του κώδικα δεοντολογίας ή χρηστών πρακτικών αν θέλετε που είχε γίνει δεκτός στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και να τον ενημερώσουμε τον κώδικα αυτό επί τη βάση των τροποποιήσεων που έχουν διαμεσολαβήσει μετά από τις νομικές αλλαγές και τις αλλαγές ε, στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Θα επανέλθει το θέμα προσυζήτηση στη συνάντηση των συντονιστών και θα καταλήξουμε νομίζω σε ένα κείμενο που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κάτι το οποίο ζητήθηκε από όλους εσάς. Γύρω από τις αιτήσει γνωμοδότησης για δύο έγγραφα, το ένα αφορά την βιοποικιλότητα και το άλλο αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας. Η σοσιαλιστική ομάδα θα αναλάβει το θέμα της βιοποικιλότητας και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το δεύτερο θέμα και θα μας ενημερώσουν σε έφετο χρόνο οι πολιτικές ομάδες για το όνομα του εισηγητή. 4 eh, Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο αναβλήθηκε για την επόμενη συνάντηση σχετικά τώρα με την ακρόαση και αυτό έχει σημασία σαν θέμα του αρμόδιου επιτρόπου σαν εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επιτροπή μας. Η συνεδρίαση των συντονιστών αποφάσισε να επιμείνει στο αίτημα και εμείς σαν Επιτροπή Αναφορών να έρθουμε σε επαφή με τον αρμόδιο επίτροπο τον αρμόδιο για τα θέματα τα οποία εντάσσονται στο δικό μας χαρτοφυλάκιο. Κάτι το οποίο είναι θα έλεγα νέο για την Επιτροπή μας η οποία ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε έναν συγκεκριμένο επίτροπο με τον οποίο να έλθει σε επαφή στο παρελθόν. Προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε έτσι ώστε να έχουμε πλέον ένα τέτοιο επίτροπο και καταφέσαμε το αίτημα αυτό όπου χρειάζεται ξεκινώντας από την διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Σας θυμίζω επίσης ότι δημιουργήθηκε και μία ιστοσελίδα για την παρακολούθηση όλων των αρμοδιοτήτων οι οποίες προβλέπονται για τον διορισμό του νέου Ombudsman. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή η σελίδα η οποία κάθε φορά λειτουργεί θα λειτουργήσει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σχετικά με την εκλογή του Ombudsman θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής στο Στρασβούργο την 19η ε, Οκτωβρίου. Θα πάρετε την πρόσκληση γύρω από την έκτακτη αυτή συνάντηση. Ελπίζω να μην άφησα τίποτα εκτός. Δεν έχει λυθεί ακόμα το τεχνικό πρόβλημα δυστυχώς. Θα ήθελε κάποιος συνάδελφος το λόγο ή μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την εξέταση των, των αναφορών και μετά να ακούσουμε τον εμπειρογνώμονα. Οπότε ας αρχίσουμε λοιπόν με τις αναφορές.

Από ό,τι φαίνεται δεν είναι συμβατό το σύστημα. Δεν βγάζει εικόνα. Ε, Θέλετε να μας κάνει την παρουσίασή σας χωρίς εικόνα. Ή να ακούσουμε πρώτα τις αναφορές μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Ερωτώ και τους τεχνικούς. Si può risolvere. same impression. Okay. Sorry, I, I, un- unless the, uh, the Εκτός και αν πρέπει να φύγει ο μιλητής, νομίζω ότι θα να ακούσουμε πρώτα μία αναφορά και μετά να επανέλθουμε. Νομίζω ότι πιο χρήσιμο θα ήταν αυτό και για τα μέλη της Επιτροπής. Αυτό θα πρότεινα λοιπόν. υπήρξε μια αντίρρηση από πλευρά τη υπηρεσία γιατί το θέμα αυτό είναι τμήμα, θα έλεγα, ενό ευρύτερου τμήματος αναφορών, τις οποίες θα ακολουθήσουμε και αμέσως μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας εξετάσουμε πρώτα τις αναφορές και μετά θα τις εμβαθύνουμε. Περνάμε στο σημείο 10 λοιπόν. Ξεκινάμε με την 251 του 2007 του Μαρίν Γκαλέα από τη Μάλτα. Θα ακούσουμε την κυρία Λορέν Κοντεφαρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, σας έλεγα. Η αναφορά αφορά καταρχάς ε, το χαρακτηρισμό ειδική ε, ζώνης προστασίας με βάση την ε, οδηγία για τα πτηνά και μια δεύτερη στην ΤΑΣΕΝΚ. Σε ό,τι αφορά την ειδική ε, προστασία, ε, αυτό αφορά τα κράτη-μέλη για το πώς θα χαρακτηρίσουν τις ζώνες και τις περιοχές ειδικής προστασίας, αλλά θα πρέπει να είναι ε, συγκεκριμένα και επιστημονικά τα κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια που αναγνωρίζουν τα περισσότερα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ένας κατάλογος που έχει ε, καταρτιστεί από το Life ε, ονομάζεται IBA, Important Bird Areas, περιοχές που έχουν σημαντική παρουσία πτηνών. Το 2004 11 ζώνες χαρακτηρίστηκαν ως ζώνες IBA, 12 ε, όρισε η Μάλτα, εκ των οποίων 10 μπαίνουν σε αυτό τον κατάλογο IBA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε μια καταγγελία και ξεκίνησε προσφυγή επιπαραλήψη και ζητάει από τις ε, αρχές της χώρας να εξηγήσουν γιατί ε, έχουν ε, χαρακτηρίσει όχι κάποιες περιοχές και ποια είναι τα επισημαντικά στοιχεία. Λάβαμε τα στοιχεία και την απάντηση της Μάλτας. Είπαμε να εφαρμόσουν το τελευταίο κατάλογο γιατί δεν μας ικανοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγήσει που έδωσαν οι μαλτεζικές αρχές. Τελικά, οι ε, επιφάνειες ε, των ε, ζωνών ΙΜΠΑ που δεν έχουν χαρακτηριστεί από τις μαλτεζικές αρχές ως ζώνες ειδικής προστασίας αντιστοιχούν κυρίως σε ζώνες ενδιάμεσες, κοντινές των προστατευμένων και είναι σημαντικές διότι είναι όχι ε, απαραίτητες ακριβώς περιοχές για τη διατήρηση των πτηνών, αλλά ως ενδιάμεσες μεταξύ ε, κατοικημένων ή ε, άλλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν είναι σε θέση να ε, απαιτήσει από τις μαλτεζικές αρχές να χαρακτηρίσουν, να αποχαρακτηρίσουν. Το άρθρο 6 της οδηγίας για τους φυσικούς οικοτόπους Habitat είναι ένα άρθρο που πρέπει να βρίσκει η εφαρμογή εδώ εκτός των περιοχών ε, του δικτύου Natura 2000. Θα πρέπει να γίνουν μελέτες επιπτώσεων και για την έγκριση και την αδειοδότηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προστασία των ειδών των πτηνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προστατεύσει την κοινοτική νομοθεσία και θα ε, είναι πάρα πολύ ε, σε Ε, τώρα, το, για το άλλο θέμα, την περιοχή του Τατσέγκ, ε, πρόκειται εδώ για την οδηγία πάλι χάπιτα των ε, φυσικών οικοτόπων. Η περιοχή αυτή θεωρείται κοινοτική σημασίας, προτάθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2008 και είναι σε ένα κατάλογο που θα εγκρίνει το Δεκέμβριο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη, γνωρίζει το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο αναφέρονται ε, οι ενδιαφερόμενοι, πρόκειται για την επέκταση υπάρχοντος ξενοδοχείου σήμερα στην περιοχή Ρατούρα 2000 και είναι και στην οδηγία Habitat και στην οδηγία για την προστασία της άγριας πανίδας και των πτηνών μάλλον. Εξ όσων γνωρίζουμε, στο έργο αυτό έγιναν ήδη πολλές τροποποιήσεις για να ε, συμμορφωθούν στην κοινοτική νομοθεσία και επίσημα θα συζητηθεί αυτό μέσα Οκτωβρίου με τις Μαλτέζικες Αρχές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει το λόγο συνάδελφοι, κύριος Μπουζουτήλ. Grazie, signora Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να θίξω είναι το εξή. Δεν καταλαβαίνω πώ η Επιτροπή αυτή μπορεί να απεστάλλει πριν από δύο χρόνια και μετά έχουμε ακόμα συζητήσει. Νομίζω ότι οι αναφέροντες θα πρέπει να λάβουν μια εξήγηση. Γιατί χρειάστηκε να περιμένουν δύο ολόκληρα χρόνια. κρατού δοθεί προσοχή στην αναφορά τους και δεν έχουν συμβεί και πολλά. Μάλλον έχουν συμβεί πολλά τα τελευταία δύο χρόνια και έχει αλλάξει η κατάσταση πλέον. Υπήρξαν εξελίξεις και σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πριν από δύο χρόνια. Μπορεί να έχει, αλλάξει, να αλλάξει η κατάσταση. Και μάλιστα, αν σωστά κατάλαβα, φαίνεται ότι όντως ε, έχουν υπάρξει εξελίξεις και η εν λόγω περιοχή έχει ανακηρυχθεί πλέον περιοχή προστατευόμενη από την οδηγία για, το, για τους οικοτόπους, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει απόφαση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δίκαιο νομίζω αυτό για του αναφέροντε. Δύο χρόνια χρειάστηκε να περιμένουν και δεν έχει ακόμα δοθεί απάντηση. Ούτε είναι σωστό προ τι ε, εταιρείε που είναι ιδιοκτήτριε ε, γη στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Άρα αυτή είναι μια δική προς όλους, προς όλες τις πλευρές. Επίσης, Πρόεδρε, να πω ότι καθόλου δεν με ικανοποιεί η απάντηση της Επιτροπής η οποία δεν είναι συγκεκριμένη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η αναφορά αυτή να τοποθετηθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει και να μας απαντήσει με σαφήνεια προκειμένου να κλείσουμε με οριστικό τρόπο την αναφορά αυτή. Θα πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Δεν μπορούμε να περιμένουν άλλο, να επιτρέψουμε να περιμένουν άλλο για αναφέροντε. Συμφωνώ. Ε, ε, ο κύριος Ατάρτ. Ατά. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφό μου για το ότι δεν ε, είμαστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί. Γιατί οι ενδείξεις είναι οι εξής. Τον Οκτώβριο θα γίνουν σχετικέ συζητήσεις για το θέμα αυτό. Για να δούμε και να σιγουρευτούμε για ποια περιοχή μιλάμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο αυτό έχει δηλώσει ότι η ανάπτυξη έχει αναδιαρθρωθεί και ότι 60% προστατεύεται ως ε, τόπος ε, εθνικής κληρονομιάς, ότι πρόκειται, όπως ξέρετε, για ιδιωτική περιουσία και ότι φυσικά θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα του τουρισμού, τα οποία φυσικά θα πρέπει να ισοσταθμιστούν με τα συμφέροντα των ε, περιοχών που προστατεύονται από το Natura. Υπό τους όρους αυτούς θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τον Δ. Μπουσουτήλ και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις τον Οκτώβριο για κάποια ζητήματα και συμφωνώ με τον δόκτωρ Μπουσουτήλ στο σημείο αυτό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβληθεί, να αναβληθεί μάλλον η αναφορά αυτή για άλλη συνεδρίαση θα είναι πιο σωστή όταν θα έχουμε δηλαδή στην διάθεσή μας και περαιτέρω στοιχεία. Αν δεν διαφωνεί κανείς, νομίζω ότι είναι σκόπιμο, συμφωνώ και εγώ, να διατηρηθεί στην ημερήσια διάταξη αυτή η αναφορά Βέβαια, να μην την αναβάλουμε επαόριστο, να τη γράψουμε στην επόμενη συνεδρίαση και στο μεταξύ να ε, έρθουμε σε επαφή και με τους αναφερόμενους για να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να λυθούν και ως προς το αντικείμενο της αναφοράς έχει περάσει πολύ καιρός και δεν είναι καθόλου αδιάφορο αυτό και άσχετο. Είναι σημαντικό. Θα πρέπει να κλείσουμε υπεύθυνα όμως αυτή την αναφορά, να ελέγξουμε τι συνέβη. Συμφωνείτε, ο συνάδελφο τη λόγη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την πρότασή σας, αλλά για να διευκρινίσουμε λίγο τα πράγματα, να πω το εξή. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα υπάρξει συνάντηση στα μέσα Οκτωβρίου με τις ε, Μαλτεζικές Αρχές, θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα και σε άλλες συναντήσεις μετά από τη συνάντηση με τις ε, Μαλτέζικες Αρχές. Άρα, να συζητήσουμε το θέμα αυτό και στην Επιτροπή μας μετά από τη συνάντηση αυτή. Μάλιστα. Καλώς, πολύ ωραία. Λοιπόν, αν δεν διαφωνεί κανείς τώρα, ας επιτρέψουμε, επιστρέψουμε ε, στην παρουσίαση. Έχουμε την τεχνική υποστήριξη πλέον. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την παρουσίαση της μελέτης. Α, τώρα δεν έχουμε ήχο. Allora, ritorniamo al punto 9, la presentazione dello studio. Eh, παρουσίαση της μελέτης, λοιπόν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Η Επιτροπή Αναφορών ε, μου ζήτησε να σας παρουσιάσω μία μελέτη που ε, ε, έγινε από μία εταιρεία συμβούλων που ονομάζεται Milieu, περιβάλλον, βάσει τη οδηγίας του Συμβουλίου 92 το 93 που έχει να κάνει με τους φυσικούς οικοτόπους, habitat. Σύντομα θα σας παρουσιάσω τα βασικά σημεία της έκθεσης. Πρέπει να σας πω ότι η μελέτη έχει ως αφετηρία μία διαπίστωση. Ότι δηλαδή συνεχώς επιδεινώνεται η διατήρηση και η προστασία των ειδών και των φυσικών οικοτόπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, όπως φαίνεται από στοιχεία επιστημονικά και από απάντηση των κοινοτικών αρχών ε, που από το 2010 θέλουν να σταματήσουν την απώλεια της βιοπικιλότητας και να δημιουργηθεί το δίκτυο φύση 2000 με συγκεκριμένα είδη που προστατεύονται ήδη από την οδηγία του 79 για την προστασία της άγριας πανίδας πτηνών και του 92 για την προστασία των φυσικών οικοτόπων. Euh, Η μελέτη που συνέταξα επικεντρώνεται βασικά στην εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας σε 8 κράτη-μέλη. Όπως γνωρίζετε, η οδηγία αυτή υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να προστατεύουν τους φυσικούς οικοτόπους που έχουν οριστεί και χαρακτηριστεί έτσι, στις διάφορες βιογεωγραφικές περιφέρειες και υπάρχουν και απαιτήσει διαδικαστικές ε, για έργα που ενδεχομένω να βλάψουν και να προκαλέσουν ζημίες σε προστατευόμενους οικοτόπους. Σύντομα θα ήθελα να θυμίσω τη δομή του άρθρου. Τέσσερα εδάφια περιέχει. Εδάφιο πρώτο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα διατήρησης και προστασίας, ιδιαίτερα συγκεκριμένα ε, σχέδια διαχείρισης. Στο δεύτερο εδάφιο υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να λάβουν ε, συμβατικές υποχρεώσεις και μέτρα για, πάλι, για πρόληψη ε, πρόκληση ζημίας ε, στις περιοχές αυτές. Το τρίτο εδάφιο αφορά την υποχρέωση των κρατών να κάνουν μελέτη επιπτώσεων αντικτύπου ε, για κάθε έργο και κάθε προγραμματισμό που σημαντικά θα επηρεάσει ενδεχομένως την περιοχή. Και το τέταρτο εδάφιο προβλέπει κάποιες παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις. όλα αυτά τα, τα έργα μπορούν ε, ενδεχομένω και σε περίπτωση ενητική να εφαρμοστούν, σε περίπτωση που πρόκειται για ψηλότερο εθνικό συμφέρον. Και επίσης το τέταρτο εδάφιο ε, μιλάει για αποζημιώσεις και μέτρα στα οποία μπορεί κανείς να προσφεύγει. Τώρα, ενεπλέξαν πολλοί σύμβουλοι για την εταιρεία Μιλιό στα διάφορα κράτη-μέλη, τα οκτώ που έγινε η μελέτη και πώς επελέγησαν τα κράτη αυτά για να γίνει όσο γίνεται καλύτερη ε, μελέτη διαφόρων περιπτώσεων. Έχουμε και χώρες από τη Δύση, από την ε, Κεντρική Ευρώπη, από το Βορρά. Όσο γίνεται περισσότερες ως δεύτερο κτίριο γεωγραφικές περιφέρειες και νομικά καθεστώτα που κυρίως είναι από το ε, ρωμαϊκό και γερμανικό δίκαιο ως προς τη φιλοσοφία των συστημάτων. Άλλο κριτήριο επιλογής. Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν οι περιοχές αυτές ε, στη συνοχή του δικτύου ε, Natura ή Φύση 2000. Να έχει γίνει μελέτη αντικτύπου περιβαλλοντικού και για το πόσο είναι σημαντικά προγράμματα. συνήθω είναι μεγάλα έργα, αυτοκινητόδρομοι, ε, έργα υποδομή και βαριές επενδύσεις. Ε, όλα τα έργα λοιπόν που συμπεριλάβαμε στη μελέτη μας ήταν επίμαχα και από οικονομική και από οικολογική και από κοινωνική πλευράς. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια λοιπόν επιλογής mm. των περιπτώσεων. Στη συνέχεια έχουμε μελέτες των εθνικών επιρογνωμόνων που αφορούν σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με θέματα περιβάλλοντος, ε, είπαμε αυτοκινητοδρόμων, φραγμάτων, ε, ορυχείων, καταστάσεις ε, ηλεκτρικές υψηλής τάσεως, μονάδες ταφής απορριμμάτων κτλ. Προσπάθησα στη συνέχεια να συγκεντρώσω αυτές τις διαπιστώσεις και να προχωρήσω σε κάποιες συστάσεις. Πρώτο, πρώτη διαπίστωση. Χαρακτηρισμοί, ε, μεγάλες καθυστερήσεις στα κρατημέλη. Πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμα το καθεστώς προστατευμένης ε, περιοχής και δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια. Αποτέλεσμα, επιδεινώνεται η διάβρωση της βιοπικιλότητας. Λοιπόν, ε, θα πρέπει το συντομότερο να ταξινομηθούν σε κατηγορίες και να χαρακτηριστούν οι περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει τα ε, καθεστώτα προστασίας, ε, τα μέτρα αυτά να αφορούν όλες τις προστατευόμενες περιοχές και να υπάρχει ξεχωριστό για κάθε περιοχή διαχειριστικό σχέδιο. Διαπίστωση δεύτερη αφορά τη φύση των εθνικών μελετών επιπτώσεων. Τι μας έδειξαν οι μελέτε στα κράτη-μέλη, ότι πολλές από τις επιστημονικές αναλύσεις δεν ήταν κατάλληλε για τους εξή λόγου. Κυρίως οι εμπειρογνώμονες δεν, δεν λαμβάνουν υπόψη τους το συρρευτικό ε, αποτέλεσμα, ε, ούτε την εναλλακτική αξιοποίηση. Δεν ήταν αρκετά, ε, πώς να το πω, εξειδικευμένοι, η η μελέτη που έγινε δεν ήταν αρκετά ε, διεπιστημονική με εξέταση διαφόρων πτυχών. Προτείνω να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη ε, όσο γίνεται περισσότερο να συμμετέχει το δημόσιο και η κοινή γνώμη, να είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και ενδεχομένως όταν ε, το έργο είναι πραγματικά επιμαχό να ζητούμε και πραγματογνωμοσύνη κατά την παράθεση. Πολλές μελέτες, και εκεί είναι το σημείο που χωλαίνει, ε, δείχνουν ότι από επιστημονικής πλευράς ε, δεν είναι πάρα πολύ στιβαρές πάντα οι μελέτες. Και εδώ έχω προχωρήσει σε κάποιες συστάσεις. Θα πρέπει οι επιπτώσεις να αξιολογούνται όχι με τρόπο φυρημένο, αλλά πολύ συγκεκριμένο. Οι έμεσες βέβαια επιπτώσεις θα πρέπει να αναλύονται και εκείνες που είναι μακροπρόθεσμες έχουν συρρευτικό αποτέλεσμα και ε, είναι μη αναστρέψιμες. Να έχουν τη δυνατότητα λοιπόν οι εμπειρογνώμονες να αναλύουν και άλλες λύσεις και άλλους τρόπους αξιοποίησης που να ε, πλήττουν λιγότερο το φυσικό οικότοπο. Έρχομαι τώρα στη λήψη των αποφάσεων. Οι περισσότεροι εθνικοί εμπειρογνώμονες μας έδειξαν, κατέδειξαν ότι ε, αγνοείται η αρχή της προφύλαξης ε, και κάτι άλλο και εδώ είναι πιο προβληματικό αυτό. Για κάποια, α, κάποιες ζώνες προτεραιότητας, ενώ η Ευρωπαϊκή Οδηγία ε, απαιτεί να γνωμοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη δεν ζητούν αυτή τη γνωμοδότηση. Επίσης, προβλέπει η οδηγία να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται όλα τα συμφέροντα. Τα κράτη-μέλη όμως τα θυσιάζουν ε, κυρίως όλα στο βωμό των οικονομικών συμφερόντων και εις βάρος της προστασίας της φύσης. Ενώ η οδηγία έχει ως κύριο στόχο την πρόθεση αυτής της διατήρησης. Ε, σας είπα ότι έχω κάνει και κάποιες συστάσεις για τη διαφάνεια και για συμμετοχή ε, των ειδικών ενδιαφερμένων. Συχνά παίρνουν ε, Αποφάσει κάποιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς να ρωτούν σε εθνικό επίπεδο κανένα ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα διατήρηση και προστασίας της φύσης. Επίσης, ζητώ καλύτερη στάθμιση των συμφερόντων και εμβάθυνση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, έτσι ώστε εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις να λαμβάνουν την απόφαση προ όφελο τη φύση ή εκείνη που είναι λιγότερο επιβλαβή για τη φύση, πάντα με την αρχή τη αναλογικότητα. Παράγραφος 4 της οδηγίας ε, προβλέπει ε, αντισταθμιστικά μέτρα, ε, παράγραφος 4 του άρθρου 6 ενώ Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κάπως απογοητευμένοι διαβάζοντας τις αναλύσεις μας, διότι τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι πάρα πολύ ευραία και καμιά φορά ανύπαρκτα. Και κυρίως εφαρμόζονται μετά το τέλος της κατασκευής του έργου, ίσως και ποτέ δηλαδή, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Και εδώ ζητώ καλύτερη εφαρμογή, πιο αυστηρή εφαρμογή στα κράτη-μέλη και μεγαλύτερη πειθαρχία. Τα αντισταθμιστικά μέτρα θα πρέπει πραγματικά να εγγυώνται τις ζημίες που έχει υποστεί η φύση. Για το δίκτυο 2000, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να γίνονται πριν την εκτέλεση και την κατασκευή του έργου για να μην έχουμε αυτές τις εξυπνακίστικες λογικές που κανένας δεν εφαρμόζει κουτοπώνυρα ε, βρών ε, τα ε, απαραίτητα μέτρα και να υπάρχουν και ε, ειδικέ κατηγορίες για μέτρα αποζημίωσης και αντισταθμιστικά. Τελευταίο, το έλεγχος. Ο έλεγχος επειδή σας έχουν βομβαρδίσει με αναφορές, όπως και το δικαστήριο παίρνει πολλές αποφάσεις για την εφαρμογή του άρθρου 6. Τα εθνικά δικαστήρια, ιδιαίτερα <clears throat> πρώτου επίπεδου, καλούνται να αποφασίσουν για τις διαφορές και νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν πυρογνωμοσύνη επιστημονική, δεν έχουν πάρα πολλά χρήματα, αντιμετωπίζουν τρομερά εμπόδια σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων τους και δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε να γίνουν οι φύλακες ενός περιπλόκου καθεστώτος. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει ένα πολύ δραστήριο ρόλο και θα συνεχίσει να διώκει τα κράτη τα οποία παραλείπουν στη βάση του 36 σύμφωνα με τη διαδικασία επί παραλήψη. Είναι θεματοφύλαξη των συνθήκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε πλήρως και αποκλειστικά αυτούς οι οποίοι φύγονται για να προστατεύουν τη σωστή εφαρμογή των νόμων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Όλα αυτά που μας είπατε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τα σχόλια που απαιτούνται, αλλά θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κρέμερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί το Κοινοβούλιο για μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη μελέτη, με την πλειοψηφία των συμπερασμάτων της οποίας είμαστε σύμφωνοι. Πράγματι το Natura 2000 και η νομοθεσία γύρω από αυτό, για τα πτηνά και για την οδηγία, οι δύο βασικές οδηγίες, είναι βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος βασική προτεραιότητα παράλληλα με την καταπολέμηση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Ε, ο αριθμός των αναφορών παραπώνων και παραβάσεων στον τομέα του Natura 2000 αντιπροσωπεύει το πέμπτο περίπου των αναφορών γύρω από το θέμα του περιβάλλοντος γενικότερα. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει το Natura 2000 και έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφυγές επί παραλήψη για καθυστερήσεις στη μεταφορά των εθνικών ομοθωσιών. Υπάρχουν 24 ανοιχτές υποθέσεις και ε, πολλές είναι ανοιχτέ σε επίπεδο δικαστηρίου. Όλα αυτά αποδεικνύουν την σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αυτά, αλλά και τη σημασία των ιδίων των θεμάτων. Γνωρίζουμε λοιπόν τη μεγάλη σημασία των οδηγιών αυτών τη μεγάλη σημασία των περιοχών Natura 2000 που είναι το βασικό μας μέσο, ένα μοναδικό μέσο σε επίπεδο παγκόσμιο θα έλεγα, αντιπροσωπεύει 25.000 τοποθεσίες οικολογικού ενδιαφέροντος και έχει σαν στόχο την διατήρηση του περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος χώρου αλλά και της πανίδας και της χλωρίδας το δίκτυο αυτό δυσκολευθήκαμε <clears throat> να μπορέσουμε να ζητήσουμε την εφαρμογή του. Μετά όμως τον εντοπισμό των τοποθεσιών, αυτή η δύσκολη φάση κλείνει. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και για το θαλάσσιο περιβάλλον και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο χαίνει είναι η σωστή διαχείριση των δικτύων αυτών όπως επίσης και η κατάλληλη χρήση ε, των μέσων που έχουμε για να πετύχουμε την εφαρμογή της οδηγίας. Εξ αρχής λοιπόν αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προσπαθεί να αναπτύξει τις κατευθυντήριες γραμμές ιδιαίτερα σχετικά με το άρθρο 6. Υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν υπάρξει πρόσφατα λεπτομερείς. Το 2007 δημοσιεύσαμε και εμείς μια ερμηνεία για το 6.3 και 6.4. Κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες για να ενισχύσουμε το διάλογο και τη συνεργασία μας με πολλούς άλλους τομείς. Να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα, σαν παράδειγμα στους λιμένες, στα δέλτα των ποταμών. Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική ομάδα εργασίας για τις περιπτώσεις αυτές έτσι ώστε επί τη βάση του 6 να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και να προωθήσουμε την ανταλλαγή χρηστών και βελτιστοποιημένων πρακτικών. Έχουμε επίσης προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για τις μονάδες παραγωγής με ολική ενέργεια, για τις εξορυκτικές δραστηριότητες και δημιουργήσαμε και μία νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση του Natura 2000, των περιοχών του Natura 2000, μια ειδική ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με θέματα προσδιορισμού των τοποθεσιών, με την εφαρμογή των προγραμμάτων διαχείρισης, με την εφαρμογή μέσων διατήρησης του περιβάλλοντος όπως προβλέπονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση και με τα νομικά θέματα τα οποία τίθενται, ξεκινήσει μια διαδικασία συνεργασίας με τους εθνικούς δικαστές για ένα πρόγραμμα σεμιναρίων. Έγινε ένα σεμινάριο στη Βουλγαρία σήμερα με πολλούς δικαστές από γειτονικέ επίσης χώρες. Θα γίνει και στη Γαλλία τον Νοέμβριο με στόχο την βελτίωση της κατανόησης και την εναρμονισμένη αντιμετώπιση της οδηγίας αυτής από τα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά στοιχεία με τα οποία συμφωνούμε από αυτά που ακούσαμε. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της ποιότητας των μελετών, διασφάλισης του ανεξάρτητου χαρακτήρα των εμπειρογνωμόνων και των καρπών της προσπάθειάς τους, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και να βλέπουμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα σε επίπεδο παραλήψεων σύμφωνα με το άρθρο 6. Αν δεν ζητηθεί η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί που είναι απαραίτητο, είναι προφανές ότι μιλάμε για μια παράληψη, παράβαση μάλλον, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει τα απαιτούμενα μέτρα. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ευχαριστώ πάντως για τη μελέτη και δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά τη μεγάλη σημασία που δίνουμε στην εφαρμογή των μέτρων γύρω από το Natura 2000. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρέμερ. Έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Χάρμα Άουκεν, Ντεμπρούν, άλλος. Άουκεν, ναι, σας είπα. Άλλος. Ωραία. Οι τέσσερις αυτοί. Η κυρία Μπελιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεσάντελερ ε, για τη μελέτη του και να υπογραμμίσω και την ποιότητα της μελέτης. Συμφωνώ ιδιαίτερως με τα συμπεράσματα. Θέλω να επιμείνω σε κάποια σημεία. Πρώτον, η πλειονότητα των αναφορών που δεχόμαστε εδώ αφορούν όντως το, την τήρηση και την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Είναι αρκετά ανισχυτικό αυτό που συμβαίνει. Το δείχνει και η έκθεση και το υπογραμμίζει η μελέτη που μας παρουσιάσατε. Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι μπορούν ακόμα και σήμερα για να παρακάμψουν τις οδηγίες αυτές και να μην τις εφαρμόσουν. Για τα άγρια πτηνά και για τους οικοτόπους δεν εφαρμόζουν την αρχή της προφύλαξης. Είτε λοιπόν στην Επιτροπή αναφορώ είτε στις μελέτες βλέπουμε ότι τα έργα σταματούν επειδή έχουν δράσει οι πολίτες και είναι το θέμα επίμαχο, υπάρχει διαμάχη ή πολιτικό πρόβλημα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Στο πεδίο εφαρμογή οδηγία για του φυσικού οικοτόπου, σήμερα, εκτό από την ανεπάρκεια πολιτική βούληση που χαρακτηρίζει τα κράτη-μέλη, έχουμε και ε, μια ελάχιστη ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν πιέζει τα κράτη-μέλη ε, να εφαρμόσουν το κοινοτικό δίκαιο. Τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω και να σας προειδοποιήσω για κάτι στην ακρόαση του κυρίου Μπαρόσο φάνηκε ότι θέλει να προτείνει αναθεώρηση της ε, οδηγίας ε, Habitat και Natura 2002. Αυτό που μας δείχνει σήμερα όμως η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι η οδηγία κύρια τάξη, αλλά η εφαρμογή της, στα κρατημέλη και ο έλεγχος αυτής. Δεν μας χρειάζονται καινούργια κείμενα. Έχουμε μηχανισμό αρκετά ευφυή και ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, συμπεριλαμβάνουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες ε, σεβόμενη τη φύση και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να εφαρμόζεται η οδηγία και ο μηχανισμός ελέγχου της. Και θα είχα και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είπαμε και γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δίκτυο Φύση ε, 2000 και γενικότερα για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ε, θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω συγκεκριμένα και με βάση τους στόχους οδηγίας για τους οικοτόπους και του μηχανισμού και τη βιοπικιλότητα. Τι γίνεται, θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση το 2010. Τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν το 2010 έτος της βιοπικιλότητας τα προηγούμενα χρόνια όλα αυτά τα προγράμματα που είχαμε δεν κατάφεραν να επιβραδύνουν την απώλεια ειδών στη φύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή. Και σε σχέση με τα εφιστάμενα κείμενα και το κοινοτικό δίκαιο, τι προβλέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπελιέ επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τζάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η εφαρμογή του Natura θα πρέπει να είναι σωστή για την προστασία των οικοτόπων και συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ότι πολλές ε, από τις αναφορές που δεχόμαστε καταδεικνύουν ότι προφανώς υπάρχει έλλειμμα στην εφαρμογή ή πολύ απλά είναι πολύ διαφορετική η αντίληψη που επικρατεί σε κάθε περιοχή για το τι θα πρέπει να γίνει βάσει κάθε νόμου. Μιλήσατε για θέματα διαχείρισης, θα πρέπει λοιπόν να τα αναφέρουμε αυτά και να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και ποιες απαιτήσει ε, θα πρέπει να πληρούνται. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι σε μεγάλα τέτοια project όπου Υπάρχει έντονη παρέμβαση στη φύση, όπου καταστρέφεται ουσιαστικά το φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή των στρωμάτων και από οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να ελέγχουμε πραγματικά το τι δημιουργούμε, τι κατασκευάζουμε. Αυτό εντάξει, αλλά θα ήθελα να θέσω και προς την Επιτροπή ένα άλλο πρόβλημα για να γίνει αποδεκτά ότι είναι όλο και λιγότερο αποδεκτά τα μέτρα ε, του Natura 2000. Δηλαδή, αν δεν προσέξουμε, θα έχουμε άλλα προβλήματα. Και στην Γερμανία αυτό αφορά ουσιαστικά δύο μέτρα, τα οποία ε, είναι πολύ αμφιλεγόμενα και στον τύπο. Το ένα είναι η απολύμανση, αν θέλετε, ε, πρώην πεδίων μάχης, πεδίων βολής, όπου υπάρχουν ε, θαμμένα ακόμα άρματα μάχης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιες όταν λέμε ότι θέλουμε πλέον να απολυμάνουμε, να καθαρίσουμε τις περιοχές αυτές και πώς εντάσσεται αυτό και στα πλαίσια του Natura και πολύ απλά θεωρώ ότι είναι δυσανάλογα τα μέτρα και ο κόσμος που ζει εκεί πέρα δεν καταλαβαίνει γιατί θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να θεωρούν δηλαδή ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες όταν πρόκειται για την απομάκρυνση των ε, αρμάτων αυτών. Ένα δεύτερο πρόβλημα ακόμα πιο ευρύ αν θέλετε στην Γερμανία, στη Σαξονία, την περιφερειά μου υπάρχουν ε, πολλές παλιές σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίες πλέον ε, έχουν παραπληστεί, δεν χρειάζονται και οι οποίες ε, με περίπλοκο τρόπο ουσιαστικά ε, θα πρέπει να αποσυρθούν. Η κοινή λογική, λογική τι λέει, ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προβλήματα, αλλά στην πράξη προκύπτουν προβλήματα βάσει του Natura 2000, γιατί χρειάζονται ε, μελέτες, ακολουθούν ε, διαμάχες ε, και καθυστερεί πολλά χρόνια η όλη διαδικασία. Είμαστε υπέρ του Natura 2000, είμαστε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο στις περιφέρειες να μην, ε, αν θέλετε, θέτουμε και διακυβεύουμε την ίδια την αξιοπιστία της νομοθεσίας μας ε, επί τόπου. Να πούμε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν σημαίνουν μεγάλη παρέμβαση και να μην ζητάμε υπερβολικά υψηλέ απαιτήσει που θα πρέπει να πληρούνται, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα γίνουν πιο αποδεκτά τα μέτρα αυτά και από τον κόσμο. Mrs. please. Η κυρία Άουκεν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω δανέζικα. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχει γίνει. Να ευχαριστήσω και κάπως πιο διστακτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί, γιατί οι εμπειρίες μου είναι αρκετά δυσάρεστες σε ό,τι αφορά την προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκπληρώσω τις ε, απαιτήσει που θέτει η οδηγία. Γιατί η οδηγία για τους οικοτόπους είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς σε ό,τι αφορά τα σχόλια και τις ενστάσεις που γίνονται για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα είναι εύκολο να μιλάμε για προβλήματα, γιατί στο σημείο αυτό διακρίνεται πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιλύει πραγματικά σημαντικά προβλήματα. Αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε και επιτόπου στον κόσμο. Και εμεί, οι πολιτικοί είμαστε υπεύθυνοι για τι εξηγήσει αυτέ για την ενημέρωση του κόσμου. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται προστασία τη φύση, γιατί θα είναι μεγάλο το τίμημα που θα κληθούμε να πληρώσουμε μακροπρόθεσμα, αν εφαρμόζουμε μόνο βραχυπρόθεσμα μέτρα. Στο Γκοτεμπορκ είχαμε πει ότι θα πρέπει να προστατευτεί η βιοπικιλότητα, να σταματήσει η υποβάθμιση της φύσης, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να τονίσω για μία φορά ακόμη ότι ήταν πραγματικά μεγάλο σοκ ο, το ότι ήρθε ο κύριος Μπαρόσο και μας είπε όταν το ρωτήσαμε για τα προβλήματα του Natura 2000 και έχουμε δει τόσα πολλά παραδείγματα αν θέλετε υποβάθμισης και επαναχώρησης και έχουμε και την έκθεση αυτή στα χέρια μας πλέον. Αναφέρθηκαν λοιπόν όλες οι λύσεις, οι εναλλακτικέ ε, λύσεις και το καθεξής, ότι η αρχή της πρόληψης και πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και μας απάντησε ότι θα πρέπει να ψωτευτούν μόνο τα πρωτεύοντα οικονομικά μέτρα. Η Κομισιόν δεν δραστηριοποιείται αρκετά στον τομέα αυτό δεν φταίνε μόνο τα κρατημέλη, φταίει και η Επιτροπή. Και μας είπε λοιπόν ο κύριος ε, Μπαρόσο ότι βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης ε, η νομοθεσία. Ναι, αλλά στην πράξη θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ελπίζω να δούμε τι ισχύει. Όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βλέπουμε όμως πόσες αναφορές υποβάλλονται και αυτό κάτι καταδεικνύει. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την δουλειά που κάνατε. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να το αφήσουμε κατά μέρος. Γιατί έχουμε συνηθίσει να τηρούμε αυτή τη στάση και στην χώρα μου. Άλλωστε και στη χώρα μου υπάρχουν τέτοιες ε, περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Όχι, εμένουμε στους στόχους που έχουν ε, τεθεί εξ αρχής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τιμπρούν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω τις ευχαριστίες μου, να ευχαριστήσω και εγώ για τη δουλειά που έχετε κάνει για την έκθεση αυτή. Μία σειρά σημείων ήθελα να θίξω. Καταρχάς το σημείο που κι εσείς ε, θίξατε με σαφήνει ότι υπάρχει όντως αποτυχία. Δεν ε, είναι έγκαιρη η προστασία των ε, οικοτόπων και δεν υπάρχουν σωστά διαχειριστικά προγράμματα για τη σωστή προστασία τους. Οι στόχοι τους οποίους θέσαμε σε ό,τι αφορά το σχέδιο των οικοτόπων και της βιοπικιλότητας. Πολύ απλά δεν πρόκειται να ε, τους πετύχουμε και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική διάσταση των οικοτόπων κατέδειξε ότι το παγκόσμιο οικονομικό κόστος για την απώλεια βιοπικιλότητας ανέρχεται σε 1,4 έως 3,4 τρισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άρα επειδή υπάρχει τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομική διάσταση και όχι στην διάσταση του περιβάλλοντος, ε, ορίστε λοιπόν ένα καλό επιχείρημα. Είναι πολύ μεγάλη η ζημία που προκαλείται και σε οικονομικό επίπεδο από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Χαίρομαι για τις ομάδες εργασίας που έχουν δραστηριοποιηθεί στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικέ βιομηχανίες, για παράδειγμα, θα ήθελα να μάθω κατά πόσο είναι σε φάση που μπορούν να δημοσιεύσουν ε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Και πότε θα συμβεί αυτό. Και ζητώ από τα κράτη-μέλη, προφανώς πρώτα από τα κράτη-μέλη, να αντιμετωπίσουν ε, τις ελλείψεις που έχει το κάθε κράτος μέλος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και θα ήθελα να αυξηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τα κάποια νέα κράτη-μέλη, στη Βουλγαρία για παράδειγμα. Έγινε μια συζήτηση και στην τελευταία συνάντηση αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Βουλγαρία και φυσικά δεν υπάρχουν δικαιολογίε για κανένα κράτος γιατί αν κάποια κράτη-μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους σύντομα, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να εκπαιδευτούν και άλλα κράτη-μέλη. Και πολλά κράτη δήλωσαν ότι χαίρονται όταν λαμβάνουν πληροφορίε που του βοηθούν να εφαρμόσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα μέτρα. Αυτό αποτελεί μόνο μία πτύχη του θέματο. και νομίζω ότι αυτό που μα αφήνει να καταδεικνύει η μελέτη είναι ότι θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά διαδικασίε εκ παραβάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί Μία πολύ βασική συνιστόσα, αλλά το γεγονό ότι από την μελέτη προκύπτει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε για την βιοπικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, σημαίνει ότι χρειάζονται πιο δραστήρια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποστινάρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή για την εξαιρετική του μελέτη. Θα συνεχίσω στη ρωμανική, σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένη οδηγίας, της οδηγίας Habitat. Υπάρχει μια σαφή σύγκρουση από, ανάμεσα στα οικονομικά συμφέροντα από τη μία και στους στόχους της συγκεκριμένης οδηγίας. Και η τουριστική βιομηχανία και οι αναπτυξιακές πολιτικές ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργούν μερικές φορές προβλήματα. Στη Ρουμανία υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αιωλική ενέργεια και για τις συνέπειες, τις επιπτώσεις των αιωλικών εγκαταστάσεων ε, στις διαδρομές των ε, πουλιών. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα βέβαια την Επιτροπή μας είναι η πάρα πολύ καθυστερημένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή εντοπιστεί ένα πρόβλημα. Όταν συζητάμε για τις επιπτώσεις ενός οικονομικού σχεδίου πάνω στο περιβάλλον, μέχρι τη στιγμή που θα ληφθεί η τελική απόφαση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ο χρόνος ο οποίος μεσολαβεί είναι πάρα πολύ μεγάλος. Από τη μία έχουμε τα κράτη-μέλη, τα οποία συνεργάζονται με ιδιαίτερους δισταγμούς, διστάζουν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ να ευνοήσουν την προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερος αργή στους ρυθμούς εργασίας της και όταν το λέω αυτό είμαι ιδιαίτερα ευγενής. Τι εννοώ αν καταλήξουμε στην διαδικασία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσφυγής επί παραλήψη εναντίον, εναντίον συγγνώμη, κράτους, στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία αυτή δικαστικά είναι post facto, για να μην πω post mortem. Είναι πάρα πολύ αργά πλέον. Η πρότασή μου συνεπώ είναι η εξή. Θα πρέπει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει σαν βασική της προτεραιότητα το εξή. Πρώτον, να διαμορφώσει μια ενιαία νομική πρακτική αντιμετώπισης όλων των κρατών μελών και να υιοθετήσει ε, συγκεκριμένες ε, πιστοποιημένες κατά κάποιο τρόπο αντιδράσεις στις ενέργειες ή στις μη ενέργειες των κρατών μελών. Γιατί αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να περιμένει χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς συγκεκριμένες προθεσμίες τις απαντήσεις των κρατών μελών. Συνεπώς τα κράτη-μέλη ε, αν δεν πιεστούν δεν πρόκειται να απαντήσουν έγκαιρα. Αν όμως οι αντιδράσεις είναι ενιαίες τότε θα μπορέσουμε να ε, βελτιώσουμε σαφέστατα ε, την εφαρμογή των οδηγιών και στη συγκεκριμένη περίπτωση της συγκεκριμένης οδηγίας Habitat για το οικοπεριβάλλον. Θα πρέπει επίσης στα πλαίσια του διαλόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες να μην αγνοήσουμε τα θέματα που άπτονται της οδηγίας Habitat. Αυτό γιατί οι συνέπειες κάποιων προβλημάτων είναι διαμεσοριακές και διασύνοριακές και σωρευτικά λειτουργούν μάλιστα. Να σας θυμίσω τι γίνεται με το πρόγραμμα για τον αγωγό Nord Stream. Ξέρετε ότι η Ρωσία έχει υπογράψει την, πρόσβα... την ε, συμφωνία, την Διεθνή Σύμβαση μάλλον για τις περιβαλλοντικές συνέπειες αλλά δεν την έχει επικυρώσει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία θα πρέπει ε, να προκληθεί κατά κάποιο τρόπο να αντιδράσει και να πάρει μέρος στις συζητήσεις που γίνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση που διαπιστούνται μη σεβασμός της ε, Οδηγία Habitat. Η Ουκρανία έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνε και για τη βιοπικιλότητα της Μαύρης Θάλασσας. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε μιλήσει για τις αρνητικές επιπτώσεις ε, ενός καναλιού που χύνεται στη Μαύρη Θάλασσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό απέναντι στην Ουκρανία. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια της Επιτροπής ε, να πάρουν μέτρα για ε, τις συζητήσεις τους με τις τρίτες χώρες. Ο κύριος Κρέμερ έχει ζητήσει πάλι το λόγο. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες τουλάχιστον. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν και προβλήματα κατανόησης ε, στην κοινή γνώμη για το τι είναι η οδηγία Habitat για τους φυσικούς οικοτόπους και ε, η φύση 2000. Στην πράξη τι σημαίνει. Έχω ακούσει επικρίσεις του τύπου ότι περιορίζονται κάποια έργα ή δυσκολεύονται κάποια έργα λόγω υπερβολικών φραγμών και εμποδίων. Μα η οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους Habitat επιτρέπει την αηφόρο ανάπτυξη, ανάπτυξη έργων υποδομής σε αρμονία με την ανάγκη προστασίας της βιοπικιλότητας. Εάν τώρα σε κάποιες περιπτώσεις, καμιά φορά η εφαρμογή, η ερμηνεία γίνεται υπερβολικά επιτόπου και ε, δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχουν ε, ε, άχρηστα εμπόδια, αυτό δεν είναι το πνεύμα της οδηγίας. Η οδηγία προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν αναπτυξιακά έργα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αντικτύπου κατάλληλη και λαμβάνεται υπόψη ε, η ανάγκη προστασίας βιοποικιλότητας. Συχνά τα έργα γίνονται με βάση τον οικονομικό σχεδιασμό. Πρώτα δηλαδή αρχίζει το έργο και μετά γίνεται η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες για τη βιοποικιλότητα. Εκεί θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Όταν προγραμματίζεται ένα έργο, τη στιγμή του σχεδιασμού του τα έργα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ένα πάρα πολύ πρώιμο στάδιο όλους αυτούς τους στόχους και τους στόχους της βιοπικιλότητας και της προστασίας. Είναι προφανές ότι αν δεν ληφθούν υπόψη αυτοί οι στόχοι από νωρί, πολύ νωρί, στο τέλος θα βρεθούμε μπροστά σε εμπόδια. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια επικοινωνία, μια ενημέρωση της κοινή γνώμη, για να έχουμε και μεγαλύτερη αποδοχή και της οδηγίας και πολύ καλύτερη λειτουργία και εφαρμογή στην πράξη. Έχουμε τις επαφές που κάνουμε ε, με τους διάφορους ενδιαφερομένους, αυτή την προσέγγιση την οποία προωθούμε, που ονομάζεται στα αγγλικά Working with Nature. Εργαζόμαστε με τη φύση. Ε, δηλαδή, προετοιμάζουμε κάποια έργα και ε, βάση του άρθρου 6.3 δεν θα πρέπει να έχουν προβλήματα στη φάση της υλοποίηση. Γιατί εκ των προτέρων από το σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πτυχέ και οι περιβαλλοντικέ και οι ανάγκη να ε, ε, ληφθούν και αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτά. Ως προς την αποδοχή και τις δυσκολίες που έχουμε σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση εκεί για τη φύση 2000. Γιατί θεωρήθηκε ότι ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια πεδία στρατιωτικών ασκήσεων ή παλιέ εντυροδρομικές γραμμέ. Όχι. Επιτρέπεται, αλλά να γίνει μελέτη και να είναι φόρο η ανάπτυξη. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι προτίθεται να ε, κάνει στο μέλλον. Οι προτεραιότητε βεβαίω είναι εφαρμοστεί το πρόγραμμα δράση για τη βιοπικιλότητα που κοινοποιήθηκε το 2006 στο Κοινοβούλιο και παρακολουθείται η εφαρμογή του και μέγιστη προτεραιότητα βεβαίω εδώ θα είναι η κατάρτιση και αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου ΦΥΣ 2000. Και όπως είπα προηγουμένως, η αποτελεσματική και συνεκτική και συνολική διαχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να παίζει ένα ρόλο ε, εκ των προτέρων να προωθεί ε, την εφαρμογή. Βέβαια από τη στιγμή που έχουμε παραβάσεις παραμένει αυτό ένα προφανές ε, στοιχείο και σύμφωνα με το άρθρο 226 προχωρούμε σε προσφυγές. Βέβαια είναι κάπως χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες. Ε, υπάρχει μια προειδοποίηση, μια ε, γνώμη στη συνέχεια τελογημένη. Υπάρχουν διαδικασίες και στάδια σε αυτή την υπόθεση η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων με τη βιοποικιλότητα, ναι, σας είπα ότι είναι συγκρόμενα συμφέροντα, αλλά η οδηγία είναι ένα εργαλείο που ε, προσφέρεται πάρα πολύ καλά για να ε, λυθούν αυτά τα προβλήματα. Αναθεώρηση της οδηγίας, αν χρειάζεται. Εμεί θεωρούμε ότι είναι μια χαρά η οδηγία. Βεβαίω είναι δύο οι οδηγίε, έτσι. Μια για την άγρια πανίδα για το 79, για τα πτηνά, και η άλλη του 92 για του οικοτόπου. Εντάξει. Ε, παράλληλα ε, εφαρμόζονται. Αν χρειάζεται αναθεώρηση, αυτό μόνο μετά από τα συμπεράσματα της ε, εφαρμογής του προγράμματα δράσης μετά το 2010 και κάποιες εκθέσεις που γίνονται για την εφαρμογή του άρθρου 17 Και μάλιστα φέτος δημοσιεύτηκε η πρώτη μελέτη και έδειξε ότι η βιοπικιλότητα κινδυνεύει, είναι σε κακή κατάσταση ακόμα. Και αν λοιπόν χρειαστεί αναθεώρηση αυτή θα γίνει για να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό αυτό το μέσο, δηλαδή για να βγουν εμ, κάποια ελαττώματα από την οδηγία αυτή και σε καμία περίπτωση για αποδυνάμωση. Δεν είναι καθόλου αυτός ο στόχος μιας ενδεχόμενης αναθεώρησης είναι το βασικό εργαλείο της κοινότητας για τη βιοπικιλότητα αυτή η οδηγία. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχουμε και χρόνο μάλλον, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Δεσάντελεύ για την παρουσίασή του. Δεν υπάρχουν άλλοι που έχουν στήσει το λόγο είναι στη διάθεσή σας ο επιδογνώμων. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. Πηγαίνουμε στις ομαδικές τώρα αναφορές, την 11. του Κάρλος Ρίος Τόρες, Ισπανού. Ο κ. Δεφαρία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Η κυρία Ντεφέρια. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξε μια προηγούμενη ανακοίνωση προς την Επιτροπή αυτή, όταν λάβαμε την αναφορά αυτή, η οποία ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικά αποδεκτικά στοιχεία. Δεν υπήρχαν επαρκείς λεπτομέρειες για το κατά πόσο υπήρχε ε, τέτοια παραβίαση για την οδηγία του οικοτόπους. Ζητήθηκαν λοιπόν επιπλέον πληροφορίες από τους αναφέροντες και ο αναφέρον απέστειλε στην Επιτροπή μια σειρά εγγράφων και έγγραφα των ε, αρχών που καταδεικνύουν ότι υπήρχε αξιολόγηση του αντικτύπου του έργου και η έγκριση που είχε χορηγηθεί για το έργο συμπεριλάμβανε μέτρα τα οποία λάμβαναν υπόψη τις ανάγκες για προστασία των ε, προστατευόμενων ειδών. Όταν απεστάλησαν αυτές οι επιπρόσθετες πληροφορίες, ο αναφέρον δεν αμφισβήτησε τις ε, Ισπανικές αρχές και άρα η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις ε, της οδηγίας για τους οικοτόπους και ότι δεν υπάρχει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ah, λοιπόν, αν κάποιος θέλει το λόγο, εάν όχι, περνάμε στο επόμενο σημείο. Αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή για να εξετάσουμε λεπτομερέστερα την απάντηση της Επιτροπής. Περνάμε λοιπόν στις 12. Στην 37-2005 την οποία κατέθεσε η Λορόνς Ντολαμαρτινιέ, Γαλλίδα. Συνέχεια της 6-13 του 2009. Είναι παρόν ο Ζω Μαρί Σαλωμό και του δίνω το λόγο για να παρουσιάσει την αναφορά του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ για τη μελέτη αυτή ως αναφερόμενος που αντιμετωπίζω μια δύσκολη κατάσταση και περιβαλλοντική απειλή. Τα συμπεράσματα της μελέτης ε, συμπίπτουν απολύτως με τις δικές μας διαπιστώσεις. Είναι πάρα πολύ καλή. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ομιλώ για τις δύο αναφορές 37 του 2005 και 613 του 2009 ως πρόεδρος ε, της Ένωσης Μαρδιεβάλ που τις ε, κατέθεσε. Επίσης θα μιλήσω εξ ονόματος των 300 πολιτών που έχουν υπογράψει κατά του έργου και ε, είμαι και η φωνή των ε, ενώσεων της Ιλίσου Λουάρ και της Μπολ που έχουμε συμμαχίσει απέναντι σε τρεις αντίστοιχες απειλές. Η αντίστασή μας ξεκίνησε και η μαρτυρία αυτό πριν από 13 χρόνια για τρεις γέφυρες επιπλέον που θέλουν να κατασκευάσουν στο ποταμό Λίγυρα. Ήδη από τον περασμένο αιώνα δεν είχαν λόγο ύπαρξης και σήμερα τελείως σε σχέση με τις διαπιστωμένε ανάγκες μιας αηφόρου βιώσιμη ανάπτυξης και λελογισμένης οικονομίας. 300 εκατομμύρια επιπλέον εκτός από το περιβαλλοντικό κόστος. Ε, η ε, περιφέρεια ε, κοινοτική της Ματιέρα από το Λουαρέα από το 1974 προστατεύεται ως πράσινη ζώνη γύρω από την πόλη της Ορλεάνης για να περιοριστεί η αστική επέκταση της ε, Ορλεάνης. Ε, είναι προστατευμένα τα δάση και ενταγμένα σε προγράμματα. Από το ΣΝΙΕΦ και ΖΙΚΟ και ε, η κοιλάδα του Λίγυρα πλέον χαρακτηρίζεται η ζώνη ειδική προστασίας στην Ατουρά 2000 από την οδηγία για τα πτηνά και κοινοτική σημασία από την οδηγία Habitat. Και από το 2000 και η κοινότητα και ο ποταμός ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Ε, έχουμε πολλά είδη σπάνια και προστατευόμενα. Πάνω από 100 ε, είδη αγρίων πτηνών. Και εκεί μπορούμε να βρούμε 40 ε, που προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάνω από 15 ιδιαίτερα εύτραυστα, όπως είναι οι ψαραετή ή τα γλαρόνια στην οδηγία αναφέρονται στο παράδειγμα 1. Οι ειδικοί βιότοποι σε ποτάμιο περιβάλλον επίσης έχουν κάστορες, ενιδρίδες, ε, οστιλαστικά ή άλλα είδη ε, αρχιπτέρων και ε, χειροπτέρων. Αρχίπτερα είναι λιβελούλη, για παράδειγμα, τέτοιου είδους ε, ε Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρόλο που είναι τεράστιος ο φυσικός πλούτος ε, και έχει διαπιστωθεί και από την Επιτροπή σας που ήρθε επιτόπου το περιβάλλον είναι ιδιαίτερου κάλους, μαγικό θα το χαρακτηρίζαμε. Παρ' όλα αυτά το Γενικό Συμβούλιο του Λούαρε το 1996 αποφάσισε να γίνει μια εκτροπή ε, για ε, τα φορτηγά, υπενώντας το Λίγυρα σε ένα μέρος που τελείως ε, ακατάλληλο είναι, 2.700 μέτρα του σημερινής γέφυρα που είναι 500 μέτρα, σε ένα έδαφος καρστικό που είναι πάρα πολύ ευτραυστό και ευαίσθητο. Δεν μπορούν να ε, δεχτούν τους 7 πυλώνες που προβλέπεται στα μείον 35 μέτρα. Αυτό σημαίνει τεράστια ε, ζημία και ενόχληση του ε, υπεδάφους. Αποφασίστηκε το έργο αυτό σαν, χωρίς να έχει ποτέ μελετηθεί καμία εναλλακτική λύση ας πούμε, θα μπορούσε η σημερινή γέφυρα που είναι και πρόσφατη να αξιοποιηθεί καλύτερα. Ο νομάρχης το είχε τότε απορρίψει αυτό το έργο γιατί δεν είχαν γίνει σοβαρές μελέτες, αλλά υποτίθεται έκτοτε έχει αιτιολογηθεί και επανειλημμένα λόγω κάποιων συγκρίσεων που έχουν γίνει, αλλά έχουμε την ε, απόδειξη ότι με κάποιες προφάσεις έχουν προχωρήσει σε στρεβλώσεις και παραχαράξεις. Ε, ε, η κοινή γνώμη επανειλημμένα με ψήφο το έχει καταψηφίσει. Αλλά οι τοπικές αρχές του νομού προσπαθούν να το σώσουν το έργο αυτό παραδίδοντάς τους ένα βαρόνο των δημοσίων έργων με μια διαδικασία ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Βλέπε νέα αναφορά του 2009, εμείς το ε, καταγγέλουμε. Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση αντικειμενική και δεν υπάρχει ενημέρωση και πρόσβαση στη δικαιοσύνη όπως πρέπει. Εγώ έρχομαι να σας καταθέσω επίσης ότι μπορεί κάποια στοιχεία της οδηγίας Natura 2000 να μην είναι αρκετά αναγκαστικά, αλλά σε αυτά βασιστήκαμε εμείς για να επικαλεστούμε ε, την προστασία της φύσης. Η ε, μελέτη επιπτώσεων για το περιβάλλον που επιβάλλουν οι οδηγίες ε, ε, απεφάνθη εις βάρος του έργου, αλλά το Γενικό Συμβούλιο το απέκρυψε αυτό για να ψηφιστεί διαφορετικά. Και τώρα σιγεί ηχθείως. Περιμένουν να το περάσουν με τη βία αυτό και αναγκαστικά. Επίσης σας λέω ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ καλό κλίμα ε, που μας επιφυλάξατε και σεβασμό. Για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, εδώ έχουμε την εντύπωση ότι μας ακούν και μας προσέχουν. Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα επιχειρήματά μας τα λαμβάνετε σοβαρά υπόψη και ισόρροπα, εφόσον πρόκειται για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ε, ρωτούν, ε, ρώτησαν οι ε, βουλευτές κάποια στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές και απαντήσαμε με ε, στοιχεία εμπεριστατωμένα και αριθμητικά. Ήρθαν οι βουλευτές και έγινε και επεισόδιο. Ε, αλλά αυτό ήρθε προς επίρρωση των όσων λέμε εμείς. Πέρασαν το λίγυρα από γέφυρες το μεσημέρι, είναι σχεδόν ε, Άδειε. Οπότε ποια είναι η συμφόρηση. Είναι ψεύδος αυτό για να χτιστεί το έργο. Να δικαιολογήσουν την αδικαιολόγητη παράκαμψη για τα φορτηγά που δεν έχει καμία αποδεδειγμένη ωφέλεια για την κοινή γνώμη. Είναι σοβαρή προειδοποίηση αυτή ε, κατά των απειλών για την παραβίαση της ε, Natura 2000. Βέβαια, ο εργολήπτης ε, προχωρήσει σε φυγή προς τα εμπρός και σε περιφρόνηση. Λάθος για μας. Να ζητήσουμε από τις αρμόδιες αρχές να αναθεωρήσουν τα έργα αυτά ε, στο Μαρδιέ. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι η Επιτροπή σα θα θα δώσει συνέχεια στα θέματα αυτά, στα αιτήματά μα και θα πιέσει τι γαλλικέ αρχές μέχρι να δικαιωθούμε ή εάν το αγνοήσουν οι αρχές αυτές θα προσφύγει ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης. Δεν θέλουμε να σας κρύψουμε, ανησυχούμε βαθύτατα για τις προθεσμίες ε, των διαδικασιών αυτών και των έργων. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κινδυνεύει τώρα να επιταχυνθεί αν περάσει στα χέρια του ιδιώτη φορέα που δεν έχει τις διοικητικές υποχρεώσεις ε, που απορρέουν από τον κώδικα για τις κατοικές προμήθειες. Τα δημόσια έργα αν θεωρήσουμε ότι είναι απλή απειλή ε, για την παραβίαση οδηγία και αυτό δεν χρειάζεται ε, τιμωρία, τι θα πρέπει να περιμένουμε να συγκεκριμενοποιηθούν, αυτό να χτιστεί η γέφυρα και μετά να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, αφού δεν το θέλουμε το έργο. Και όταν ε, οι ε, ζημιές που έχουμε προβλέψει δυστυχώ θα είναι ανεπανόρθωτες, ήδη μα έχουν κόψει το δρόμο προ τη διοικητική δικαιοσύνη τη Γαλλία, λέγοντα υποτίθεται ότι δεν έχουν ε, χαρακτήρα λήψης απόφασης αυτές οι υποτιθέμενες ε, απειλές. Μα υπάρχει σύμβαση του άρχους που είναι κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούν να μας αρνούνται την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Υποχρεούνται τα κράτη σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και των σωματείων και των ενώσεών τους. Δέκα χρόνια μετά την κύρωσή της η Γαλλία δεν έχει αλλάξει ούτε κατά ένα κόμμα αυτή τη διαδικασία. Και ε, με τη δική μας αναφορά 613 του 209 που ευχαριστούμε που την κάνετε παραδεκτή. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή την κατάσταση. Το Γενικό Συμβούλιο, από ό,τι φαίνεται, ε, θα ανοίξει τα σχήρες του γιατί δίνει την εργολαβία σε ένα ιδιώτη στα πλαίσια μιας ΔΙΤ, σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Στη δική μας υπόθεση, το Γενικό Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου του 2009 ενέκρινε 106 εκατομμύρια ευρώ για ε, το σχέδιο αυτό του Μαρτιέ ε, στις ΔΙΤ αυτό το έκανε αγνοώντας την υποχρέωση που είχε να αποδείξει ότι δεν υπήρχε πιο φτηνή εναλλακτική ικανοποιητική λύση. Δεν υπάρχει καμία ε, απάντηση, όλα τα έχουν αφήσει στις ορέξεις των ε, ιδιωτών για τις τέσσερις γέφυρες δεν υπάρχει κανένα σεβασμός, καμία αιτιολόγηση, ε, δεν λαμβάνονται υπόψη ε, τα συμπεράσματα της μελέτης για το Natura 2000 που χωρίς καμία αμφισημία έλεγαν ότι δεν ε, υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτή η γέφυρα στο Μαρτιέ. Η χρηματοδότηση, η ψηφοφορία για τη χρηματοδότηση λοιπόν δεν είναι μια απόφαση λιμένη που ε, παραβιάζει την οδηγία. Δεν θα έπρεπε η ίδια Ευρώπη να αναθεωρήσει τις πρακτικές της για να ε, συμμορφωθεί με τη σύμβαση του Άρχους και να μην περιμένει ε, να επιβεβαιωθούν τα λάθη και να έχουμε φτάσει σε καταστάσεις ανεπανόρθωτες. Έχουμε τώρα ακόμα καιρό. Η Επιτροπή Αναφορών θέλησε να μας υποστηρίξει, ήταν αποφασιστικό και παραμένει για τη συνέχεια για μας αποφασιστικό και ε, σας ε, είμαστε ευγνώμονες βαθύτατα. Ε, στη Γαλλία έγινε η διαδικασία για το περιβάλλον, η συζήτηση αυτή, το γκρενέλ του περιβάλλοντος. Ακολούθησε νομοθεσία για να ζούμε με τρόπο πιο αηφόρο και βιώσιμο να αναπτυσσόμαστε, να σεβόμαστε και να σώσουμε τη βιοπικιλότητα. Ε, όλα αυτά είναι αξιέπαινα, αλλά εάν υπάρχουν και άλλες ολιγορίες, τελικά θα γίνει το έργο και με βάση τη λογική της ε, ανάπτυξης, μια λογική όμως του παρελθόντος. Η πραγματικότητα καταρρύπτει όλους αυτούς τους μύθους ότι χρειάζεται δίθεν παράκαμψη. Μόνο τα κοινοτικά όργανα λοιπόν, τα θεσμικά όργανα έχουν την απαραίτητη απόσταση από την κατάσταση για να επιβάλλουν την προστασία που ε, απορρέει από τις οδηγίες έτσι ώστε ο Λίγυρας να μην υποστεί άχρηστες και μη ε, αντιστρεπτές ε, καταστροφές. Τώρα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να περάσουμε στα έργα. Θα πρέπει αυτή η κακή περιπέτεια το συντομότερο να τερματιστεί χωρίς ε, περισσότερες ζημιές και χωρίς περισσότερες πατάλες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα την άποψη της Κομισιόν, ο Ντέβιντ Γκριμό, για την Εκτελεστική Επιτροπή. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Κύριοι αναφερόμενοι, σα ευχαριστώ μου δίνετε την ευκαιρία να σας δώσω κάποιες, κάποια στοιχεία ενημέρωσης για αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, η Κομισιόν έχει παρακολουθήσει από πολύ κοντά το θέμα αυτό και έχουμε παρέμβει πολλές φορές στην Επιτροπή Αναφορών για να δώσουμε μία ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη στο θέμα αυτό. Οι τελευταίες πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τις γαλλικές αρχές και έχουν ως εξής. Μεταξύ των σχεδίων για τις γέφυρες, μεταξύ των οποίων και τις γέφυρες του Ζαργκό, δεν υπάρχει καμία έγκριση που έχει δοθεί για την ε, κατασκευή αυτού του γεφυριού. Αυτό σημαίνει δεν έχουν περατωθεί ακόμα οι μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου βάσει της Natura 2000 και θα είναι έτοιμες μάλλον το Σεπτέμβριο 2010 και οι συμπληρωματικές μελέτες για τα θέματα περιβάλλοντος μετά από την παρέμβαση της Επιτροπής Αναφορών που ζήτησε να εξεταστεί το σωρευτικό αποτέλεσμα των ε, γεφυρών που έχουν κατασκευαστεί στο Λίγυρα δεν έχει ακόμα περατωθεί αυτή η διαδικασία. Λέτε λοιπόν ότι έχει αποφασιστεί το σχέδιο αυτό, έχει αποφασιστεί από το Γενικό Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα η πλήρης έγκρισή του. Χρειάζεται μία ε, έγκριση από τον τοπικό νομάρχη για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό υπάρχει πάντα η δυνατότητα του κοινού να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης απόφασης. Έχουμε δύο οδηγίες που είναι πολύ σημαντικές για το θέμα αυτό. Την 85 η οποία έχει στη συνέχεια τροποποιηθεί και επίσης την οδηγία 92-43 που είναι γνωστή και ως οδηγία Αμπιτά. Βάσει λοιπόν της προηγούμενης οδηγίας που ανέφερα, της 85-35, πρέπει να υπάρχει πάντα πληροφόρηση του κοινού βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα 4 όταν και εάν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Είναι οι πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν το σχέδιο, τον αντίκτυπο που θα προκύψει για το περιβάλλον από την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, περιλαμβάνονται επίσης τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και αναφέρει ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις. Σήμερα, βάσει των πληροφοριών των γαλλικών αρχών, δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Είμαστε ακόμα στα πλαίσια της ε, εκπόνησης της μελέτης αντικτύπου στο περιβάλλον. Οι τοπικές λοιπόν αρχές και οι αρχές του νομού αυτού του δεπατεμό έχουν φυσικά τις προθέσεις να κάνουν οδοποιία, κατασκευή γεφυριών κτλ. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι τα σχέδια αυτά θα γίνουν πραγματικότητα εκτός εάν οι δημόσιες αρχές δώσουν την έγκριση που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση αυτών των υποδομών και βρισκόμαστε ακόμα μακριά από αυτό το χρονικό σημείο. Οι γαλλικές αρχές είπαν ότι πριν από τον ε, Ιανουάριο του 2011 δεν θα ζητηθεί καν η έγκριση για αυτήν την ε, κατασκευή. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, έχει την πρόθεση να ζητήσει από τις γαλλικές αρχές μία περαιτέρω ενημέρωση για την κατάσταση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά την ε, σχέση αυτή, τη σύμπραξη ιδιωτικής και δημόσιας πρωτοβουλίας, ιδιωτικού και δημοσίου, ε, δημόσιων φορέων. Ο συνάδελφός μου ίσως μπορεί να σας περιγράψει περισσότερα στοιχεία για τη μορφή αυτής της σύμπραξης η οποία προβλέπεται. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον από τις γαλλικές αρχές είναι ότι δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα αυτή η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου για την ε, δημιουργία αυτού του γεφύρ, αυτού, αυτής, αυτής της γέφυρας. Αυτή λοιπόν η εταιρική σχέση θα υπόκειται και αυτή σε μία διαδικασία έγκρισης που θα ακολουθηθεί από τη διαδικασία έγκρισης της κατασκευής της γέφυρας αυτής. Δηλαδή, εάν υπάρχει αυτή η απόφαση να δοθεί ο κατάλληλος προϋπολογισμός, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσει η σύμπραξη αυτή, αλλά πρέπει να υπάρξει και η έγκριση για την κατασκευή του γεφυριού. Πάντως, μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας προβλέπεται μια δημόσια ε, έρευνα, ώστε μέσα στα πλαίσια αυτής της έρευνας οποιοδήποτε πολίτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αντικτύπου και η Κομισιό θα παρακολουθήσει από πολύ κοντά αυτήν τη διαδικασία και εμείς θα ζητήσουμε από τις γαλλικές αρχές να μας διαβιβάσουν όλες αυτές τις μελετές βαστού Natura 2000 τις μελέτες αντικτύπου στο περιβάλλον, τις συμπληρωματικές μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε, όπως απαιτεί η οδηγία Habitat, ότι κανένα σχέδιο το οποίο έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, σε συγκεκριμένη περίπτωση στην περιοχή του Λίγυρα, δεν θα μπορέσει να γίνει χωρίς την απαραίτητη έγκριση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σερβένε θέλει να λάβει το λόγο ή αν είναι επαρκής η παρέμβαση του εκπροσώπου της Κομισιόν, του προηγούμενου εκπροσώπου της Κομισιόν. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θέλω να δώσω τρεις διευκρινήσει σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν στα πλαίσια της δεύτερης αυτής ε, αναφοράς της 613-2009 και που έχει να κάνει με την ρύθμιση για τη σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την κατασκευή της γέφυρας του Μαντιέ. Πρόκειται λοιπόν για την σχέση τη συμβατική που θα πρέπει να συναυθεί μεταξύ μια ιδιωτική επιχείρηση και του δημόσιου τομέα. Αυτέ οι διαδικασίε δεν καλύπτονται γενικά από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η συμφωνία σύμπραξης η οποία προβλέπεται στην περίπτωση αυτή είναι μια συμφωνία η οποία καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από την Εθνική Ένωμη Τάξη της Γαλλίας ακόμα και αν υπάρχει κάποια ε, παραπομπή, κάποια αναφορά για τις συνθήκες ε, ε, απονομής του των διαγωνισμών στην κοινοτική νομοθεσία. Επομένως δεν υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στραφεί κατά της, ε, των δημοσίων αρχών της Γαλλίας σε σχέση με το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως την επιλογή του αντισυμβαλόμενου, του εργολάβου, υπάρχουν κάποιες διατάξεις ευρωπαϊκές οι οποίες αναφέρονται και στην ε, αναφορά και το Γενικό Συμβούλιο του Δεπατμόν του Λουαρέ ανεξάρτητα από την ε, επιλογή του θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα τρίτο φορέα για να εφαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με τους δημόσιους διαγωνισμούς. Δεν βρισκόμαστε όμως όπως ελέγξει στο σημείο αυτό. Η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρος και μακροσκελής και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ποιος θα είναι ο παρτενέας στον ιδιωτικό τομέα, η ιδιωτική αυτή επιχείρηση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι λοιπόν η ιδιωτική επιχείρηση η οποία θα αναλάβει αυτή την εταιρική σχέση με το Γενικό Συμβούλιο του Λουαρέ και επομένω η συμφωνία για τη σύμπραξη θα μπορέσει να γίνει μονάχα μετά τη διαδικασία επιλογή, η οποία είναι μια μακρά διαδικασία και η οποία μπορεί να είναι ανταγωνιστική αν πληρούνται ορισμένε προ, προδιαγραφέ για την ε, της και τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υπάρχουν λοιπόν σε όλη τη διάρκεια αυτή τη διαδικασία οι δυνατότητε να υπάρξει προσφυγή πριν από την υπογραφή του της τελικής σύμβασης. Από τη στιγμή βέβαια που συνάπτεται η τελική σύμβαση είναι πολύ δύσκολο να ανακόψει κάποιο κάποιος αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει όμως ένα σύνολο κοινοτικών ε, ρητρών και δυνατοτήτων προσφυγής κατά μιας ενδεχόμενης συμφωνίας και προβλέπεται μια σειρά υποχρεώσεων των δημοσίων αρχών για να είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το συμφέρον που μπορεί να έχει κάποιος να δράσει στην περίπτωση της ε, ε, απόφασης Λάρους φυσικά έχει περιοριστεί η έννοια του ένομου συμφέροντος με το οποίο μπορεί κανείς να παρεμβεί σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά σίγουρα το θέμα του περιβάλλοντος παίζει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο φάκελο αυτό και αν υπάρξει κάποια διαδικασία, αν υπάρξει κάποια, κάποιος ο οποίος θα καταδείξει ότι η διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού δεν θα έχει τηρηθεί σωστά, εμείς είμαστε φυσικά έτοιμοι να παρέμβουμε ενώπιον των γαλλικών αρχών για να σου υποδείξουμε ότι πρέπει να πράξουν άλλα σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ και πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Εγώ θα σας πρότεινα να περάσουμε στο σημείο 13 που είναι η αναφορά 551 καθώς 2008 του Ολιβιέ Περαιών και είναι παρόν ο κύριος Κολόν και επίσης και ο κύριος Jean-Paul Declerc ο οποίος είναι πρόεδρος της ε, Ένωσης που, ανα, που ασχολείται για τα θέματα αυτά. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους αναφερόμενους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Νταβίρ Σολό. Είμαι άλλα το παραγωγός και εκπροσωπώ τους εργαζόμενους στις Αλικές και τους παραγωγούς στην ε, περιοχή αυτή των Ελών της Γκεραντ. Σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι δεχτήκατε να εξετάσετε την ε, αναφορά μας και μας έχετε προσκαλέσει να την παρουσιάσουμε. Πρόκειται για μια κατασκευή στα όρια του έλους της Γκέραντ. Ο ωκεανός και η ιστορία έχουν δημιουργήσει τις πιο νότιες αλικές της Ευρώπης σε έκταση 2.000 εκταρίων που καλύπτει 9 δήμους. Το έργο του Αλατορίχου είναι μία από τις ε, λίγες αγροτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιεί μία τεχνική η οποία παραμένει χειρονακτική και παραδοσιακή. Και με τον τρόπο αυτό δεν έχουμε τους ίδιους κινδύνους ρήπανσης όπως και στις βιομηχανικές δραστηριότητες. Δεν παράγουμε μονάχα αλάτι. Με τη δράση μας ανανεώνουμε το περιβάλλον των αλικών και διατηρούμε και ένα φυσικό και πολιτιστικό ε, κληροδότημα και διατηρούμε τις βάσεις μιας αηφόρου ανάπτυξης. Η προστασία αυτού του φυσικού περιβάλλον είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της εργασίας μας και για την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης και επίσης και για τη διατήρηση παραγωγής ενός άλατος το οποίο είναι διεθνούς φήμης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με την εργασία μας δημιουργούμε μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή μας που αντιπροσωπεύει 450 άμεσες θέσεις εργασίας και έχει γενικό τζίρο 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χωρίς να υπολογίσουμε τις Ελκόμενε ελκόμενες από αυτή τη δραστηριότητα άλλες απασχολήσεις που είναι σημαντικές για την περιοχή μας. Η περιοχή μας αυτή έχει θυγεί από τις ε, πράξεις ορισμένων οι οποίοι θέλουν να κάνουν αστική ανάπτυξη στην περιοχή αυτή. Εμείς βλέπουμε να υπάρχει διάβρωση συστηματικά της περιοχής του φυσικού αυτού χώρου των αλικών που έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου μόνο το 70% των αλικών είναι σε κατάσταση εκμετάλλευσης. Ο κύριος Ζωάν Πολ Πολλοί τοπικοί εκλεγμένοι θεωρούν ότι οι φυσικές περιοχές είναι περιοχές οι οποίες πρέπει εν καιρό να κτιστούν. Και αυτό είναι τελείως αντίθετο και με τις ίδιες αρχές της Natura 2000, διότι με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπουν την προστασία του ε, τοπικού περιβάλλοντος το γήπεδο αυτό για το οποίο ο Δήμαρχος της Γκεράντ έχει δώσει άδεια κατασκευής, άδεια οικοδόμησης, βρίσκεται σε ένα νησί όπου από, από το, του οποίου η περιοχή τροφοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος, τα δύο τρίτα, το ένα τρίτο μάρον του έλους το οποίο είναι αλατοφόρο. Και το νησί αυτό διασχίζεται από μια συνδρομική γραμμή η οποία ήδη έχει οδηγήσει σε πρώτες κατασκευές κοντά στην θάλασσα. Δίνοντας λοιπόν μια τέτοια άδεια οικοδόμησης στην περιοχή που φαίνεται κόκκινη στην ε, αεροφωτογραφία 2, ο δήμαρχος της Γκεραντ θέλει να συνεχίσει την διαδικασία οικοδόμησης σε μια περιοχή που τη θεωρεί παρθένα και χωρίς καμία χρήση. Παρ' όλα αυτά, αυτό το γήπεδο βρίσκεται σε μια περιοχή προστατευόμενη και ιδιαίτερα ε, ευαίσθητη, η οποία έχει καταταγή στην κατηγορία ZPS στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φυσικών Χώρων της Natura 2000. Όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες, ο δήμαρχος της Γκεραντ γνώριζε ήδη από τις 13 Σεπτεμβρίου 2005 και χωρίς καμία απόλυτη αμφιβολία και ήδη προηγουμένως ότι το εν λόγω γήπεδο ήταν στην περιοχή η οποία προβλεπόταν να παραμείνει εν προστασία. Το γεγονός ότι η απόφαση η υπουργική για τον καθορισμό αυτής της περιοχής ήλθε μετά από την ε, απόδοση της άδεια κατασκευής 30 Μαρτίου 2006 μας καταδεικνύει ότι δεν υπήρξε δυνατότητα να αντισταθούμε σε αυτή την απόφαση. Στις 9 ε, Δεκεμβρίου 2005 λοιπόν υπεγράφει αυτή η άδεια οικοδόμησης για το σχέδιο Βενεσί, Βενετία, που αναφέρεται και ως ε, το αγρόκτημα του καζίνου. Με τον τρόπο αυτό όμως ο δήμαρχος της Γεράντ έχει παραβιάσει την οδηγία 9243 της 21ης Μαΐου 1992. Το να δοθεί αδεια οικοδόμηση σε περιοχές αλικών και ελών οι οποίες είναι προστατευόμενες αυτό αντιτίθεται στην Natura 2000. Μια τέτοια λοιπόν ε, κατασκευή στα όρια των προστατευμένων περιοχών ήδη αντιβαίνει σε οποιοδήποτε στόχο προστασίας των περιοχών αυτών. Εξάλλου, θεωρούμε ότι το Διοικητικό Δικαστήριο της ΝΑΝΤ, στο οποίο προσέφυγε η Ένωσή μας, όταν αποφάσισε ότι ο Δήμαρχος δεν παρεβίασε την οδηγία 92-43 δεν έλαβε υπόψη στοιχεία ευρωπαϊκού δικαίου τα οποία οπωσδήποτε θα έπρεπε να είχε πράξει ως εθνικός δικαστής. Θεωρούμε επίσης ότι ο αρμόδιος υπουργό, παρά την παρέμβαση της Ένωσής μας δεν έκανε το καθήκον του να εφαρμόσει την οδηγία αυτή αρνούμενος να γνωμοδοτήσει με το πρόσχημα ότι η υπόθεση αυτή εκκρεμούσε ενώπιον των δικαστηρίων. Θεωρούμε τέλος ότι το γαλλικό κράτος αναμένοντας το 2006 για να καθορίσει την περίμετρο της Natura 2000 στην περιοχή αυτή έχει ε, κάνει ένα σημαντικό σφάλμα αφήνοντας τη δυνατότητα στους ε, εργολάβους, στους, στις οικοδομικές εταιρείες να φτιάξουν σχέδια τα οποία παραβιάζουν αυτήν την τόσο εύθραυστη ζώνη. Είναι παρα, πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι απόψεις αλλάζουν. Μέσα στα πλαίσια του καθορισμού της περιμέτρου Natura 2000, το γαλλικό κράτος διατηρεί την ε, ταξινόμηση αυτής της περιοχής μέσα στην περίμετρο του Natura 2000 και ποτέ δεν ανετράπει αυτό από την Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για το σχέδιο Natura 2000. Λοιπόν, υπάρχει ομόφωνη άποψη ότι αυτή η περιοχή δεν θα πρέπει να τύχει κατασκευών. Θέλουμε επίσης να αναφέρουμε ότι ο Δήμος της περιοχής έχει δημιουργήσει ένα σχέδιο για την ε, αποκατάσταση των, απο, των ε, μη χρησιμοποιουμένων αλικών στην ίδια αυτή περιοχή. Μετά από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές έχει εκλεγεί νέος δήμαρχος στην περιοχή της Γκεράντ. Αυτός μπορεί να έχει μια πιο κριτική στάση έναντι του σχεδίου αυτού και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι θεωρούν ότι ήταν εσφάλματο να δοθεί η άδεια κατασκευή στην περιοχή, η οικονομική άδεια. Εξάλλου, το Γενικό Συμβούλιο έχει αγοράσει ένα τμήμα αυτή τη περιοχή, αυτού του γηπέδου, για να εξασφαλίσει τη διατήρηση του φυσικού του χαρακτήρα. Δεν έχουν κατασκευαστεί οι κατοικίε οι οποίε προβλεπόταν, αλλά θέλουμε να σα υπενθυμίσουμε ότι είναι απαραίτητο να τονιστεί προ τι γαλλικέ αρχέ ότι για να σεβαστούν την ε, οδηγία Natura 2000 θα πρέπει να δημιουργήσουν σαφή περίμετρο για τα, τις περιοχές Natura 2000 και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περατωθεί η τρέχουσα αυτή κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα ε, θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Τζόζεφ Φαντερστέγεν. Ah. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι, κύριε Κιμό, θα ε, ήθελα ε, να σας πω ότι θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Γκριμό και μετά θα συνεχίσω εγώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι αναφερόμενοι. Μιλώ για την αναφορά αυτή για να ορίσω και να συγκεκριμενοποιήσουμε το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται εδώ όπως πολύ σωστά θύμισαν οι αναφερόμενοι, το χρονοδιάγραμμα ανάμεσα στην έκδοση της οικοδομικής αδείας και τη διεύρυνση της μέτρου της προστατευόμενης ζώνης είναι σημαντικό το χρονοδιάγραμμα. Διότι διαπιστώνεται ότι πριν ληφθεί η υπουργική απόφαση εξεδόθη άδεια. Δηλαδή υπήρχε η οικοδομική άδεια και στη συνέχεια λήφθη υπουργική απόφαση που διεύρυνε το περίμετρο. Τη μέρα έκδοσης αδείας το συγκεκριμένο έργο δεν ήταν στην προστατευόμενη περιοχή, αλλά σε μια περιοχή που θα εντασσόταν αργότερα στο σχέδιο για τις προστατευμένες. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν όντως, ε, με βάση το γαλλικό δίκαιο αυτό λέγεται ζήκο, που είναι ορνοθρολογικού ενδιαφέροντος. Λοιπόν, με βάση αυτή την νομοθεσία δεν μπορεί κανείς να χτίσει ό,τι θέλει εκεί. Υπάρχει η νομολογία που λέει το άρθρο 6 ε, με βάση ε, την οδηγία Άμπιτα δεν εφαρμόζεται, αλλά ε, η παράγραφος 4 για την οδηγία για την άγρια πανίδα για τα πτηνά. Και τι λέει το άρθρο 4 παράγραφος 4, ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγουν στις προστατευόμενες περιοχές που θα έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί τέτοια, τα μέτρα λοιπόν που προλαμβάνουν τη ρήπανση, την καταστροφή των οικοτόπων και τη διαταραχή της ζωής των πτηνών. και διαταράσσεται σημαντικά ο στόχος της οδηγίας. Αυτό λοιπόν το άρθρο 4.4 για την προστασία είναι πιο περιοριστικό από το άλλο άρθρο της Habitat, το 6.2 και 6.3. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα εδώ να εγκριθεί ένα έργο που έχει σημαντικό αντίκτυπο ε, στην ζώνη αυτή. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω και να θυμίσω το νομικό πλαίσιο που ισχύει. Ο συνάδελφος μου τώρα, Βαντεστέκεν, θα σας πει τα τεχνικά του ζητήματος. Voilà, donc, je vais poursuivre. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω εγώ. Ναι. Έγινε ε, συνεδρίαση με τις αρμόδιες αρχές στις 6 Φεβρουαρίου 2009 στο Παρίσι και οι γαλλικές αρχές μας έδωσαν μια σειρά στοιχείων που είχαμε ζητήσει. Μας έδωσαν το καλοκαίρι αυτά τα στοιχεία, δηλαδή ε, αντίγραφο της οικοδομικής αδείας, ε, έκθεση στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, του νομού του, του, νομού, του ενδιαφερόμενου τις ε, νομαρχιακές αποφάσεις με το χαρακτηρισμό ε, για τα υδρολογικά, μελέτη για την Πανίδα και τη Χλωρίδα του Ιουλίου του 2007, μετά την έγκριση και χορήγηση της οικοδομικής αδείας και επίσης ε, τις υδρολογικές μελέτες και την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Νάντης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν έλαβε τη γνωμοδότηση του 2006 της τοπικής περιβαλλοντικής υπηρεσίας ούτε τα χαρακτηριστικά του νέου έργου, διότι άλλαξε το έργο έκτοτε. Από την αρχή του δηλαδή έχει εξελιχθεί. Ε, πάρα πολύ σύντομα θα στείλουμε επιστολή στις γαλλικές αρχές για να μας δώσουν τη γνωμοδότηση της περιφερειακής ε, διεύθυνση περιβάλλοντος, νομαρχιακής μάλλον, ε, στοιχεία που δεν έχουμε ακόμα. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αν το σχέδιο αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις με βάση την οδηγία για τα πτηνά. Θα ενημερώσει την Επιτροπή σας, η Επιτροπή για τα συμπεράσματα της ανάλυση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπελέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά τα δύο θέματα για να υποστηρίξω και να προσθέσω και μερικά στοιχεία για τα πραγματικά γεγονότα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο φάκελο για την περίπτωση των αλικών της Γκεράουντ, εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να συμμεριστώ την νομική ανάλυση της Κομισιόν για το νομικό πλαίσιο αυτής της υπόθεσης. Νομίζω ότι έχουμε πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία προβλέπει ότι όταν ένα κράτος έχει αμελήσει τις ε, υποχρεώσεις του βάση του κοινοτικού δικαίου, ιδίως το να καθορίσει τις περιοχές της Natura 2000 όπως θα έπρεπε, δεν μπορεί να κρύπτεται πίσω από αυτήν την παράληψη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το γεγονός ότι δόθηκε η άδεια οικοδόμησης πριν από τον καθορισμό της περιοχής ε, ως ZPS, τη στιγμή που θα, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει με μεγάλη ευκολία πέντε χρόνια από την απόδοση της άδεια οικοδομικού χαρακτήρα, αυτό αποτελεί μια σαφή και κατάδυλη ε, έλλειψη κανονικότητας από την πλευρά του γαλλικού κράτους. Αυτά σε ό,τι αφορά τα νομικά θέματα. Έρχομαι τώρα στο τεχνικό επίπεδο. Μας λέει η Κομισιόν ότι δεν έχει πάρει ακόμα την τελευταία ε, γνωμοδότηση από τις γαλλικές αρχές που έχουν ε, που έχει αρμοδιότητα στα θέματα περιβάλλοντος και ότι έχει αποσταλεί αλληλογραφία προς την κατεύθυνση αυτή στην τοπική κυβέρνηση, στις τοπικές αρχές να. Το γεγονός τώρα ότι από πολιτική άποψη υπήρχε η δυνατότητα βάσει των νέων στοιχείων και της προόδου των γνώσεων για το θέμα αυτό, νομίζω ότι εδώ το... η συναπτώμενη φωτογραφία 2 καταδεικνύει το ότι υπάρχει μια σημαντική, ένα σημαντικός ρόλος της περιοχής αυτής που αναφέρεται σε σχέση με την περιοχή προστασίας των αλικών. Δεν είναι η φύση η οποία λοιπόν στρέφεται κατά της οικονομικής δραστηριότητας. Η φύση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Νομίζω λοιπόν ότι αν δούμε συνολικά τα στοιχεία του φακέλου, εγώ θα ήθελα να κάνω μια πρόταση προς την ε, Εκτελεστική Επιτροπή και, και στην πρόεδρο της ε, Επιτροπής μας θα ήταν ίσως χρήσιμο να υπενθυμίσουμε κυρία Πρόεδρε εξ ονόματος της Επιτροπής μας να στείλουμε μια επιστολή στον νέο δήμαρχο, ο οποίος και αυτός περιμένει κάποιο νεύμα από τη δική μας περίπτωση, για να σταματήσει αυτό το σχέδιο το οποίο ξεκίνησε από κάποιον άλλο δήμαρχο. Να στείλουμε λοιπόν ένα, μια επιστολή στον δήμαρχο και στον Υπουργό περιβάλλοντος, ώστε να εκφράσουμε την βαθύτατη ανησυχία μας σε σχέση με το σχέδιο αυτό και το σημαντικό αντίκτυπο που θα έχει τόσο σε νομικό όσο και σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Αυτά αφορούσαν τον πρώτο φάκελο. Για το δεύτερο φάκελο τώρα... για την <clears throat> επέκταση του οδικού δικτύου στο διαμέσμα του Λουαρέ. Εδώ έχω μια πολύ μεγάλη δυσκολία για να κατανοήσω το περιεχόμενο αυτού του φακέλου. Η εντύπωση που έχω είναι ότι οι γαλλικές αρχές σε διάφορα επίπεδα αρμοδιοτήτων παίζουν κρυφτούλι μαζί μας από το 1996, εδώ και πάρα από 10 χρόνια δηλαδή. Υπάρχει ένα σύνολο σχεδίων. Αν δούμε το χάρτη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη παράκαμψη οδική της πόλης της Ορλεάνης, που ουσιαστικά θα επιτρέπει την ταχύτερη διάβαση από τα αυτοκίνητα οχήματα, όλο αυτό θα μπορούσε να είχε παρουσιαστεί με έναν τρόπο ο οποίος θα ήταν πιο συνεκτικός και πιο σαφής και έτσι θα είχαμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και να ζυγίσουμε καλύτερα τα θετικά στοιχεία αυτού του σχεδίου έναντι των ε, μειονεκτημάτων του. Αλλά εδώ βλέπουμε ένα κατακαιρματισμό του σχεδίου για να αποφύγουμε ακριβώ μια τέτοια συνολική ε, ε, αποτίμηση και λήψη απόφαση. Έχουμε λοιπόν ένα κρυφτούλι, έχουμε μια απόφαση που παίρνεται εδώ, μια που δεν παίρνεται εκεί. Σιγά σιγά λοιπόν δεν λαμβάνονται κατακαιρματισμένα αποφάσει σε ένα σημείο σε ένα άλλο και δεν έχουμε μια συνολική εικόνα για το φάκελο αυτό. Βάσει λοιπόν των τελευταίων στοιχείων που έχουμε, δεν είναι εκπληκτικό ότι ανησυχούν οι αναφερόμενοι για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση ενός σχεδίου ήδη έχει προβλεφθεί, έχει ξεκινήσει ουσιαστικά το σχέδιο τη στιγμή που δεν έχει δοθεί η απαραίτητη άδεια από τις δημόσιες αρχές. Υπάρχει λοιπόν απόλυτη αδιαφάνεια σε σχέση με τον φάκελο αυτό. Και αντί να περιμένουμε να υπάρξουν αποφάσεις όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο αναφερόμενος <clears throat> θα πρέπει να καταφύγει στη δικαιοσύνη, στην εθνική δικαιοσύνη και η Κομισιόν θα πρέπει να φέρει τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράληψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Natura 2000 και της προστασίας της βιοποικιλότητας, εγώ θα ήθελα να προτείνω στην Κομισιόν και στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή να δράσουμε προληπτικά στέλνοντας αυτή την επιστολή προς τις τοπικές αρχές και προς τον ε, αρμόδιο Υπουργό για την Οικολογία για να εξηγήσουμε ποιες είναι οι ανησυχίες μας και να τονίσουμε ότι πέραν των ανησυχιών μας αυτά τα οποία τεκταίνονται στην περιοχή είναι πράγματι μη φυσιολογικά σε ό,τι αφορά την προστασία της, ε, του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα λάβω υπόψη τις αιτήσει σας και εγώ θα ζητήσω από τις αρμόδες αρχές να μας απαντήσουν. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Γκρούνη Ζητώντα τη να είναι πιο σύντομη. Ζητώ από του διερμηνείς να παρατείνουμε για πέντε λεπτά ακόμα, αλλά πρέπει να κλείσουμε και θα επανέλθουμε το απόγευμα. Κύριε Γκρούν. Θα είμαι σύντομη. Για τη δεύτερη αναφορά, για τη Γεράντα, θα ήθελα να σας πω ότι έχω εκπλαγεί πολύ από τη διαδικασία αυτή. Από πλευράς νομικής δεν τα βρίσκω σωστά αυτά. Ακριβώς. Ε, πολύ συγκεκριμένα και πολύ γρήγορα θα ήθελα να ε, παρέμβουμε και ε, να κάνουμε διάβημα και στο νέο Δήμαρχο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε την απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στους αναφερομένους, γιατί πάει καιρός. Και βεβαίως υπάρχει και το περιβαλλοντικό σκέλος, αλλά και το οικονομικό εδώ. Και στη Γαλλία Μα αρέσει πολύ το αλάτι της Γεράντ. Και ε, φυσικά είναι και εκπληκτικό το τοπίο και θα πρέπει να σωθεί και γρήγορα να δοθεί Άκουσα αυτά που λέει η κυρία Μπελιέ. <laughs> Αλλά δεν έχουμε αρκετά στοιχεία πιστεύω στη διάθεσή μας. Δεν υπάρχουν μελέτες επιπτώσεων. και δεν μπορώ να αποφανθώ εγώ αυτή τη στιγμή. Και καλό θα ήταν να απαντήσει η Γαλλική Δημοκρατία για ε, τα ζητήματα αυτά που αφορούν ε, τους αναφερομένους και τους αναφερομένους. Ευχαριστώ. C'è ancora un intervento Έχουμε και άλλη παρέμβαση. Σύντομα. Σύντομα είπαμε. Γιατί πίεσε και ο χρόνος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να απαντήσω εν συντομία στην αξιότιμο κυρία Βουλευτή. Το νομικό πλαίσιο. Ακριβώς επειδή τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να κάνουν ό,τι τους κατέβει στις περιοχές που έχουν καθοριστεί περιοχές Natura 2000, το άρθρο 4 και όχι το άρθρο 3 που είναι πιο εύκαμπτο σε ό,τι αφορά την προστασία των περιοχών που είναι βιότοποι πτηνών πρέπει να εφαρμοστεί. Και αναφέρεται στο γεγονό ότι πρέπει να υπάρξει σημαντική βλάβη στον βιότοπο ή στα φυσικά είδη που προστατεύονται από την οδηγία. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να εξασφαλίσουμε το κατά πόσο το σχέδιο αυτό έχει τη δυνατότητα να έχει τέτοιο σημαντικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να προβλεφθούν για να μειωθεί ή για να εξαλειφθεί αυτός ο δυνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο έχουμε ένα πρόβλημα πράγματι. Και θα υπάρχει πραγματικά μία περίπτωση μη σεβασμού του άρθρου 4 παραγράφου 4. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 3. Πάντω τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να κάνουν τι θέλουν και εμείς εφαρμόζουμε όλες αυτές τις ρήτρε που έχετε αναφέρει. Και επίσης για να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο θέσατε για το θέμα της Ορλεάνης, έχουμε μια διαδικασία στη Γαλλία όπου ζητούμε να μας δώσουν τα στοιχεία των μελετών που έχουν, που έχουν εκπονηθεί μέχρι τώρα, να ζητήσουμε ποια, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρισκόμαστε. Επομένως, διατηρούμε επαφή με τις γαλλικές αρχές, κάνουμε